Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασης. ...18 Φεβρουαρίου, όχι 17 όπως είπα. Έχουμε μια σειρά από ψηφοφορίες και θα ξεκινήσουμε έτσι την ημερήσια διάταξη. Είμαστε σε αυτή την αίθουσα εδώ που είναι κάπως ε, διαφορετική. Θα ήθελα στην αρχή να κάνουμε μια ψηφοφορία ελέγχου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Δυστυχώς δεν έχουμε οθόνες εδώ για να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ξεκινάει τώρα λοιπόν μια ψηφοφορία ελέγχου. Άρχεται.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 Fine. Then... Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την έκθεση Μαρινέσκου. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία μπορείτε να τη διαβάσετε μπροστά σας υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία. Όχι, οπότε ψηφίζουμε την 11 όπως τροποποιείται. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική 2 και τροπολογία 15 ενστάσεις, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία 15 όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 Περ. κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά ελέγχουμε την τροπολογία 16 άρχιτη ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Αφού εγκρίνεται η 16 κατά 17 συνεχίζουμε 18 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Καταπίπτει, συγγνώμη. 23 καταπίπτει επειδή εγκρίθηκε 24. Ευχαριστώ. Ε, τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Συμβαστική 4, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής 4. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 35 έρχεται ψηφοφορία 35 όχι 34 έχουμε μία ψήφο του ΕΛΚ παραπάνω Ένα παραπάνω του ΕΛΚ. Ωραία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. «36 με προφορική τροπολογία 3». Έχει κάποιο ένσταση για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 36 λοιπόν όπως τροποποιήθηκε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ και 43 είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 45. Συμβαστική 6, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ,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 όχι, η 56 απορρίφθηκε, Συνεπώ πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία 57. Ξεκινάει λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 57. Ψήφισαν άπαντες, τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 68 τη ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 68 Συνεχίζουμε με την 69 και 70. ίδιες ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 Ένσταση όχι. Ψηφίζουμε την 72 λοιπόν όπως τροποποιήθηκε προφορικά. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές επαναλαμβάνουμε για την 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, εγκριθεί 85, 86 και 87 καταπίπτουν. Δεν εγκρίθηκε 85, συνεπώς 86 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ας τσεκάρουμε την 86. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ηλεκτρονική ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πέραμε τώρα στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ΕΚΟΝ, ΕΚΟΝ 2 όποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΕΚΟΝ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έκον 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι κάποιος κατά της μαζικής ψηφοφορίας. Όχι. Ας ψηφίσουμε λοιπόν μαζικά όλες τις τροπολογίες έκον από την 5 μέχρι το τέλος όποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, επί του συνόλου της έκθεσης ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Γκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινέσκου. Τον κύριο Σίγητη, ευχαριστούμε πολύ. I continue the votes. Συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες με την έκθεση Μπαλτσίτης.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 αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα μπορούσαμε από το 15 έως το 17 να ψηφίσουμε όλες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 18 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται, ναι. περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, προφορική, κανείς δεν είναι κατά, 12 όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δύο σημείο ακόμα. Έμπλ 1 και 2. Να ψηφίσουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ για τις δύο της Επιτροπής Απασχόλησης. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία υπέρ μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι τέλος της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια κύριε Μπαλτσίτης. Yep. Um, Μόλις μου λένε ότι πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας, υπάρχει ο νέος κανόνας που πέρασε με το ελεγκτικό συνέδριο και συνεχίζουμε με την έκθεση της κυρίας Γκρέσλε. Η ένα και οι δύο είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέντε και έξι. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελέγχουμε την 5 και 6. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Υιοθετούνται. 4. Καταπίπτει. 4. 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική για την 11 είναι κάποιος κατά όχι ψηφίζουμε λοιπόν την 11 όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ Α, συγγνώμη, καλύπτεται αυτή. Προφορική του εισηγητή, της εισηγήτρια, συγγνώμη. Είναι κάποιος κατά. Δεν μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε, είστε κατά. Συνεχίζω με την 21, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, όχι, 21, ποιος είναι υπέρ, ξαναψηφίζουμε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 με ψηφοφορία σε τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Αρχή. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Συνεχίζουμε. Αν υιοθετηθεί 23, καταπίπτει, όμως μόνο ένα τμήμα της 23 υιοθετήθηκε. Τι κάνουμε με αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν και θα δούμε κατόπιν. 22 υπέρ. Ψηφίζουμε κατά αποχές. Απορρίπτεται 22. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 κατά τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 καλύπτεται. Συμβαστική 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Α, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επανέρχομαι στην 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Όχι, επίτητες το είπα, για να τον κοιμάστε. 30. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εννοείται ότι απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 με προφορική τροπολογία. Όχι, αποσύρεται χωρίς λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ χωρίς προφορική τροπολογία. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία χωρίς την προφορική για την τροπολογία 33. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 13 κατά. 34 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά. Αποχές, Απορρίπτεται. Σαράντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζω 39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38. Δεν καλύπτεται από τη συμβαστική 8, μάλλον καλύπτεται. Συμβαστική 6, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 44, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τη 45. 46, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Α, δεν ψηφίζουμε. Ίσως θα ήταν καλύτερα να ψηφίσουμε πρώτα την συμβιβαστική. Ναι, 48, 49, ταυτότητες υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία 48 και 49. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος εγκρίνονται. Συμβιβαστική 7, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52, 53, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, 52 και 53. Αρχή της ψηφοφορίας, ψηφίσατε όλοι, Τέλος. Όντως δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται 13 υπέρ, 13 κατά. Προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος κατά. Όχι, ψηφίζουμε. 52, 53. Δεν εγκρίθηκαν, αποερήφθησαν οι 53-53. Προφορική τροπολογία λοιπόν υπέρ, κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή. Ψηφίσατε όλοι απαξάπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. υπέρ. Υπέρ της 54. Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11α με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 έχει αποσυρθεί συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 56 εκπίπτει συνολική ψηφοφορία στο σύνολο της έκθεσης άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρασε 21.4.1. Συγχαίρω την κυρία Γκρέσλε για την πάρα πολύ σημαντική αυτή έκθεση για το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Mr. Okay. Dear colleagues, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω την προσοχή σας λιγάκι. Έχουμε μια τροποποίηση της ημέρας διάταξης για τεχνικούς λόγους γιατί για το σημείο 19 ο κύριος ε, Καταλήν δεν έχει έρθει ακόμα. Έρχεται με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο εδώ στο Κοινοβούλιο, οπότε το θέμα αυτό ε, θα πρέπει να το καθυστερήσουμε και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ρούμπικ, ο οποίος συμφωνεί να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Ε, γιατί και ο υπεύθυνο του ελεκτικού συνεδρίου για τα άλλα σημεία δεν είναι παρόν και περνάμε για αυτό το λόγο, και το σημείο 20 δεν είναι παρόν, και γι' αυτό προτάσουμε το σημείο της ημέρησιας διάταξης 52, το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το απόγευμα. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίρρηση και δίνω το λόγο στον κύριο Ρίμπιχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ομοιόμορφη αλλά και όχι ιδιαίτερα θετική πάντα. Υπάρχει μεγάλη ανεργία σε, πολλά, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη να μπορέσει να προωθήσει τη βιομηχανική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις μας και θα πρέπει να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της σε ε, παγκόσμιο επίπεδο η Ευρώπη και αυτό μπορεί να γίνει κυρίως με παραγωγή νέων προϊόντων και παροχή νέων υπηρεσιών ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν ευκαιρίες για να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη παρουσία στο διεθνή οικονομικό χώρο. Με το σχέδιο 2020, το οποίο ακολουθεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, έχουμε θέσει νέους στόχους και ένα νέο πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια περικοπή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε επιτύχει το πρόγραμμα Horizon 2020 να προσαρμοστεί στις ε, ανάγκες οι οποίες αναφέρονται. Έχει εξασφαλίσει το Κοινοβούλιο ότι θα δοθούν ε, ποσά τα οποία κανονικά προβλεπόταν να είναι 100 δισεκατομμύρια από το Κοινοβούλιο, από τα κράτη-μέλη το μείωσα για το επόμενο αυτό διάστημα σε 80 δισεκατομμύρια και έχουμε προγράμματα όπως το Artemis το οποίο έχει να κάνει με τα ενσωματωμένα πληροφορικά συστήματα αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αεροναυπηγική και τη διαστημική βιομηχανία με την οποία ε, είναι ιδιαίτερα ενεργή σε θέματα σε, με εταιρείε όπως το Airbus. Υπάρχουν εταιρείε όπως η ENIAC που είναι ιδιαίτερα σε καλή θέση για τα νανοτεχνολογικά στοιχεία των υπολογιστών και των ενσωματωμένων συστημάτων. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα η Ευρώπη να ανακτήσει την, ε, ε, εξέχουσα, την προεξάχουσα θέση της στους τομείς αυτούς και έχουμε επίσης τα συστήματα FCA, την χρήση υδρογόνου στις μεταφορές. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορέσουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μεταβούμε από τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα σε νέες μορφές ε, καυσίμων και σε νέες μορφές χρησιμοποιώντας ε, υδρογόνο και ηλεκτροκίνηση και τα λοιπά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υπάρξουν ηλεκτρονικά ε, συστήματα τα οποία θα μπορέσουν να ελέγχουν αυτές τις νέες μορφές κίνησης και επομένως όλα αυτά είναι κεντρικά στοιχεία της τεχνολογικής αυτής ε, προόδου. Πιστεύω λοιπόν ότι στο επερχόμενο χρονικό διάστημα θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο γιατί έχουν ένα καινοτόμο χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για τα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία μπορούν να έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην ε, περίθαλψη στο μέλλον και έχουν αποδείξει σε μεγάλο βαθμό την αξία τους ήδη στον ερευνητικό τομέα. Μπορούμε λοιπόν με μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών να εξασφαλίσουμε ένα μεγαλύτερο ρόλο της ε, έρευνας και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα αναπροσανατολίσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επίσης έχουμε το πρόγραμμα για την θερμοποιητική σύνδεξη, το γνωστό ITER, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι με αυτό μπορούν να προκύψουν τεχνοβλαστοί, spin-offs. Υπάρχουν πολλά τεχνολογικά επιτέγματα τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερο ε, πεδίο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εφαρμοστούν στην παραγωγή. Ξέρουμε λοιπόν ότι το Διεθνές Αυτό Consortium, το ΙΤΕΡ, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα με τη χρηματοδότησή του, αλλά πιστεύω ότι οι διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να τηρηθούν και θα πρέπει να αναπτύξουμε ορισμένες κέρυες τεχνολογίες, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος στα θέματα αυτά. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα CESAR για την ασφάλεια στους ανοιχτούς εθέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να κάνει με, την, με, τον, έναρχο, με τον έλεγχο της ε, εναέριας κυκλοφορίας με στόχο να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση του εναέριου χώρου και να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων από τα αεροσκάφη. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι στοιχεία που συνάπτονται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων συστημάτων. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά να τα λάβουμε υπόψη το Δεκέμβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του 2014 μπόρεσα να πάρω μια προσωπικά να πάρω μια ιδέα για τα διάφορα αυτά προγράμματα, ε, τα επισκέφτηκα προσωπικά, άκουσα και συζήτησα με τους υπευθύνους για τις νέες αυτές δυνατότητες για τα νέα για τις κοινέ αυτές ερευνητικές δραστηριότητες και ξέρουμε και από το ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν υπήρξε κάποια αρνητική γνωμοδότηση. Μετά από όλα αυτά δεν νομίζω ότι χωρεί κάποιος λόγος για να μη δεχθεί το Κοινοβούλιο να δώσει την ε, απαλλαγή για όλες αυτές τις κοινέ ερευνητικές ενέργειες. Υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα με ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία δεν ήταν σε θέση να συγχρηματοδοτήσουν αυτές τις ενέργειες, αλλά έχουμε... Έχουμε συζητήσει για τα θέματα επίσης ιδιαίτερα των καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι <clears throat> μετά από τις συζητήσεις που έχουν γίνει και με το ελεκτικό συνέδριο υπήρξε και η σημαντική συμβολή του ελεκτικού συνεδρίου διότι δεν περιορίστηκε μονάχα στο να να ελέγξει όλες αυτές τις κοινέ ενέργειες αλλά έπαιξε και ρόλο συμβούλου για να τις υποστηρίξει. Ο στόχος εδώ είναι να μειωθεί το επίπεδο των σφαλμάτων και αυτό δεν είναι θέμα μονάχα ελέγχου, είναι απαραίτητο να υπάρξει και η απαραίτητη κατάρτιση και μετεκπαίδευση των ειδικών υπαλλήλων του ελεκτικού συνεδρίου που είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο που έχει κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες για τα θέματα αυτά που απέβησαν θετικές προσπάθειες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είδαμε ότι με τον τρόπο αυτό μπόρεσε να μειωθεί ο ο όγκος των σφαλμάτων, το ποσοστό των σφαλμάτων και συγχρόνως κατέστη δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και επομένως μετά από όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε την απαλλαγή για όλες αυτές τις κοινέ ε, ενέργειες στον ερευνητικό τομέα και να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάλει σε αυτή τη ε, διαδικασία απαλλαγής. vielen Dank äh, an den Berichterstatter. Ευχαριστούμε τον Παουλ Ρούμπιχ, τον εισηγητή. Έχετε κάποιες ε, παρατηρήσεις, θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Η κυρία Γκρέσλε. Να ευχαριστήσω απλώς τον εισηγητή. Και ήταν σωστό να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ αποκεντρωμένων φορέων και κοινών ενεργειών που ξεκίνησαν ε, πρόσφατα και επομένως υπήρχε μια ανάγκη ε, μαθητείας και κατάρτισης της κοινέ ενέργειας. Ε, ξέρουμε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι η απόφαση στην οποία ε, καταλήγουμε ήταν ιδιαίτερα θετική. Και ξέρουμε και όπως είπε και το ελεκτικό συνέδριο ότι τα αρχικά προβλήματα έχουν ξεπεραστεί και βελτιούται η κατάσταση. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις εκθέσεις, που... για τις εκθέσεις του και να εκφράσω τη συμφωνία μου με τη χορήγηση επαλλαγή στι κοινέ επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεν πρέπει να επαναπευόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη βελτίωση. Περαιτέρω βήματα θα πρέπει να γίνουν ιδιαίτερα για τη διασφάλιση μια πιο πειθαρχημένη δημοσιονομική διαχείριση δεδομένων και των αντίστοιχων προσπαθειών που γίνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται σωστά με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή να εξεταστούν διεξοδικά οι κοινέ επιχειρήσει σε μια ξεχωριστή έκθεση δεδομένων των σημαντικών ποσών που διακυδεύονται και των κινδύνων που υπάρχουν σε αυτέ τι επιχειρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει να πάρει το λόγο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτά τα κοινά εγχειρήματα, κοινέ επιχειρήσεις είναι ένα πολύ καλό πρότυπο έτσι ώστε οι σχέσεις ε, μεταξύ του δημόσιου τομέα και των, ε, του ιδιωτικού στο μέλλον να βοηθήσουν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που σήμερα γνωρίζουν η ευρωπαϊκή οικονομία. Όλοι ξέρουν ότι ο τομέας της έρευνας επιστήμης πρέπει να υποστηριχθεί και ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Υπογραμμίζω εδώ ότι ίσως ε, στο μέλλον θα ήταν λογικό να συνεχίσει η δημιουργία τέτοιων κοινών εγχειρημάτων Νομίζω ότι και για τον κόσμο της έρευνας ε, δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο νέες θέσεις απασχόλησης, προσελκύονται ε, νέοι και φυσικά είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμες τέτοιου είδους επενδύσεις. Πρόεδρος, δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο της ημέρης της διάδοξης. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τώρα αναρωτιέμαι. Μπορούμε να συνεχίσουμε και με ποια έκθεση. Εν τω μεταξύ, ο εισηγητή για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει έρθει. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Βλέπω ότι ξεπεράσατε τα προβλήματα κυκλοφορίας που αντιμετωπίσατε ερχόμενος από το αεροδρόμιο. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο που αφορά την απαραγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για το σημείο 19. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένα. Όσον αφορά την λογοέκθεση Όπως ε, μπορείτε να κατανοήσετε πιθανότατα είναι μια έκθεση ιδιαίτερης ευαισθησίας ε, όσον αφορά τη συνολικότερη απαλλαγή για την τρέχουσα ε, θητεία. Μιλάμε για τη διαχείριση των οικονομικών Συγγνώμη, κάποιες γλώσσες λείπουν από τη διερμηνία. Έχουμε μόνο τα αγγλικά, αλλά όχι τα γερμανικά. Κύριε Σιγητή. Μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά, συγγνώμη που σας διακόψα. Λοιπόν, πρόκειται εδώ για μια έκθεση ιδιαίτερης ευαισθησίας. Είναι η πιο ευαίσθητη ίσως ε, από όλη τη δέσμη των απαλλαγών, διότι Βρισκόμαστε δύο βήματα πριν τις εκλογές και μιλάμε εδώ για τι δημοσιονομικές απαλλαγέ για την οικονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου το 2012. Αυτό φυσικά είναι το θέμα μας, αλλά το θέμα αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης των δημοσιονομικών από το Κοινοβούλιο. Πρέπει να παραμείνουμε επαγγελματίε αντικειμενικοί και να μην τα τρέψουμε ε, αυτές τις εκθέσεις σε ένα προεκλογικό μέσο Καλό λοιπόν είναι που διεξάγεται η συζήτηση αυτή ουδέτερα και επαγγελματικά και με διαφάνεια. Όπω γνωρίζετε, στην εκθέση προτείνουμε την απαλλαγή, τη η απαλλαγή για το Κοινοβούλιο και λάβουμε αυτή την απόφαση αφού μελετήσαμε του λογαριασμού, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και πιστεύω ότι με την ανάγνωση των εγγράφων αυτών μπορούμε να χορηγήσουμε την απαλλαγή. Θα έλεγα ότι το πρώτο σημείο αναφορά σε αυτή την άσκηση αναφέρεται στην ε, άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου των εξωτερικών και των αυτόνομων ελεγκτών που συνάδει με την ε, άποψη των εσωτερικών ελεγκτών. Το ελεγκτικό συνέδριο στις αξιολογήσεις του δηλώνει ότι το ποσοστό σφάλματος ε, είναι σχεδόν μηδενικό και οι διοικητικές δαπάνες πραγματοποιούνται αποτελεσματικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν το 2011 να ακολουθήσουν μια οικονομική πολιτική χαρακτηρισμένη από εξοικονόμηση χρημάτων. Έτσι πράξαμε το 2011 και το 2012. Καταφέραμε λοιπόν να εξοικονομήσουμε χρήματα όπως είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε εννοείται ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό χωρίς να αποδυναμωθεί αυτή η τάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ή άλλως είναι ένας μοναδικός οργανισμός στον κόσμο. Το θέμα των εδρών είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα συνεπώς, αλλά αυτό θα εξαρτεί από τις αποφάσεις των κρατών μελών. Στην έκθεση αυτή συμπεριλάβαμε τις μελέτες ανάλυσης του προβλήματος των τριών εδρών. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε το Κοινοβούλιο για τις δαπάνες που σχετίζονται με τις τρεις έδρες αφού η αποφάσεις εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη σε κάθε περίπτωση. Επίσης με την προσοχή στις δαπάνες για τα ακίνητα και τη συντηρήσή τους. Υπογραμμίσαμε το θέμα αυτό και αναφέρουμε ότι δεν πρέπει πρέπει να ξεχνάμε αυτή την πτυχή όταν γίνονται νέες δεσμεύσεις για κινητά από το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις δαπάνες ασφαλείας ε, για εμάς και για τα κτίρια θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα μέσω του δικού μας προσωπικού για αυτή την ασφάλεια. Είναι σημαντική η ασφάλεια των προσώπων, των κτίριων αλλά και η κυβερνοασφάλεια. ασφάλεια. Πρόσφατα γίναμε στόχος ε, επιθέσεων στο διαδίκτυο. Ξέρουμε ότι πρέπει να προσέχουμε και το ζήτημα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη μελέτη που θα μας δίνει τα πραγματικά στοιχεία του κατά πόσο είμαστε στόχος τέτοιων κυβερνών επιθέσεων κατά πώ θα είμαστε τέτοιο στόχο στο μέλλον και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα ύψιστα επίπεδα ασφάλειας ε, από αυτή την άποψη στο μέλλον. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τη εκθεσή μου. Αναμένω τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ιβαν για την εκθεσή σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ο κύριος Δε πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον εισηγητή. Υπάρχουν κάποια κάπως ασαφή σημεία εδώ για την ε, διαδικασία, υπήρχαν μάλλον για τη διαδικασία του 2011 και είχα ζητήσει να λάβει χώρα μια συζήτηση και κλεισμένο το θηρό για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα για τις ε, ε, πληρωμές που αφορούν τις αποδοχές του προσωπικού. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το τι θα γίνει σε σχέση και με το 2012. Θέλω να έλθω στο θέμα αυτό και να ακούσω και την άποψη Γενικής Γραμματείας του Κοινοβουλίου αλλά ξέρω ότι θα κατατεθούν κάποιες τροπολογίες με στόχο να διευκρινιστούν καλύτερα τα σημεία αυτά για την έλλειψη διαφάνειας που αφορά την διαδικασία αυτή απαλλαγή και θα υπάρξουν και κάποιες τροπολογίες σε σχέση με την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις, ε, στους προκυρισόμενους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Δημόσιους Διαγωνισμούς και επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που θα αναφέρουν οι τροπολογίες αυτές σε σχέση με το κόστος της μετακίνησης του Κοινοβουλίου και της διασποράς του σε τρεις έδρες. Και εξακολουθώ να έχω κάποια σχόλια ακόμα για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, για το Europal, την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί ζητήσαμε να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες από τους υπευθύνους σε σχέση με την απαλλαγή του έτους 2010 στο παρελθόν και πήραμε απλώς μια γενική <clears throat> εικόνα αλλά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά. Γενικά όμως είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπικ και η κυρία Γκρέσλε ζητάνε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση. Όσον αφορά εδώ το θέμα του ελεγκτικού των κοσμητόρων, συγγνώμη, Έχω συμπετάσει σε αυτήν την απαλλαγή, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιες διαμαρτυρίες ή παράπονα των ευρωβουλευτών καλό θα είναι να ληφθούν υπόψη από τους κοσμήτορες. Και αν είχαμε εδώ μια έκθεση για το πού υπάρχουν προβλήματα, θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε τις πιο σωστές λύσεις. Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι που μπορούμε να το ζητήσουμε. Ο Αντιπρόεδρος που είναι υπεύθυνος για το τμήμα αυτό θα ήταν καλό να πάρων και επαναλαμβάνω οι αποφάσεις που παίρνουμε εδώ θα έπρεπε ίσως να έχουν ληφθεί υπόψη. Ο αρμόδιος ε, αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας θα μπορούσε να επιληφθεί του θέματος αυτού. Ίσως λοιπόν για όλους εμάς αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά σημεία. 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές και εκτός ε, συναντώνται άτομα εδώ σε αυτά τα κτίρια, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα λοιπόν της υγείας είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, να υπάρχουν τακτικοί έλεγχοι, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία για τις ασθένειες και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα για τους συνεργάτες μας, επειδή όπως ξέρετε είμαστε υπεύθυνοι, επειδή υπάρχει μία συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη, θα θέλαμε να ξέρουμε, εκτός από τη μέτρηση της θερμοκρασίας, να γίνεται και ένας έλεγχος της ποιότητας του αέρα, παραδείγματος χάρη μέσα στα κτίρια στα οποία εργαζόμαστε. Υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχει εδώ ένα ε, πρόγραμμα ελέγχων ιατρικών ε, εξετάσεων γιατί πραγματικά υπάρχουν κάποιες επαναλαμβανόμενες ασθένειες και ελπίζω να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος της και εισηγήτρης της κυρίας Ότης. Δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πρόκειται για μια, θα έλεγα, πολύ γλυκιά, ομαλή έκθεση όσον αφορά τις διαπιστώσεις της και βεβαίως ε, κάποια σημεία κατά κάποιο τρόπο προσιάζονται με σχετικά ομαλό τρόπο. Ε, είναι όντως ε, ευαίσθητο το θέμα, δεν είναι εύκολο κάποιος να αντιμετωπίσει με πιο αυστηρό τρόπο κάτι που τον αφορά εδώ δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει όμως από εκεί και πέρα και ένα θέμα αξιοπιστίας των προτάσεων και των διαπιστώσεων μας. Παραδείγματος χάριν, όσον αφορά το θέμα του mobbing, των μαζεμάτων για τα προηγούμενα χρόνια κάθε φορά διαπιστώνουμε με λύπη αυτά τα φαινομένα. Εδώ δεν βλέπω καμία αυστηρότητα όσον αφορά τις ε, διαπιστώσεις. Το θέμα της έδρας των πολλών εδρών, παράγραφος 51, το οποίο εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφές ότι υπάρχει μία έδρα στη Στρασβούργο. Απλώς υπάρχουν πολλοί τόποι στους οποίους εργάζεται το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να διορθωθεί η διατύπωση. Το θέμα της ασφάλειας, της νέας γενικής διεύθυνσης. Εδώ θα θέλαμε λίγο περισσότερα στοιχεία, λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Πολλές αποφάσεις έχουν ληφθεί από αυτήν την νέα γενική διεύθυνση. Και εδώ όλα αυτά υπάρχουν στο σημείο 12. Η Γενική Διεύθυνση Communication. Εδώ στο σημείο αυτό αναφέρεται και όλα τα ποσά τα οποία έχουν ε, δοθεί και μου φαίνεται εντελώς παράλογη αυτή εδώ η χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος και υπάρχουν και αντικρώμενα συμφέροντα. Με κανένα λογικό τρόπο δεν βλέπω να έχει αναλυθεί και παρουσιαστεί εδώ εξάλλου υπάρχει και μια τροπολογία που αφορά αυτά τα 80 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις και θα ήθελα να υπάρξει μια πραγματική δήλωση για τα ποσά αυτά, να ξέρουμε δηλαδή ακριβώς πώς διατέθηκαν εδώ πρόκειται πραγματικά για ποσά τα οποία ξεπερνούν κατά πάρα πολύ, είναι 60 εκατομμύρια ευρώ και ξεπερνούν κατά πάρα πολύ αυτά τα οποία δίνονται παραδείγματο χάρη κατά μέσο όρο στη Γερμανία για αντίστοιχε δραστηριότητε. Και πραγματικά σας λέω, εάν δίνονται αυτά τα ποσά για την ε, εκλογική εκστρατεία, σε σύγκριση με ποδιά, με τα ποσά που δίνουμε στη Γερμανία, πραγματικά είναι υπερβολικά. Εδώ πραγματικά θα ήταν πολύ καλύτερο να υπήρχε μια καλύτερη προετοιμασία και καλύτερες λύσεις για τέτοιου είδους προβλήματα. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να, είμαστε, να μην είμαστε αμερόληπτοι σε μια τέτοια έκθεση που μας αφορά. Εδώ πλήττεται η αξιοπιστία μας και το λέω με μεγάλη σαφήνεια η αμεροληψία εδώ είναι πραγματικά απαραίτητη. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Υπάρχουν τρόποι να γίνουν έξυπνες περικοπές και υπάρχουν προτάσεις. Ήδη στην περσινή ετήσια έκθεση είχαμε υπογραμμίσει κάποιους τέτοιους τομείς. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε κανείς να συνδυάσει τις δύο εκθέσεις για να υπάρχει κάποια συνέχεια στις περσινές προτάσεις. Εγώ και επ' αυτού θα κάνω κάποιες τροπολογίες. Συμφωνούμε λοιπόν με αυτά που διαπιστώνει ο συγητής. Το θέμα είναι πώς μπορούν να βρεθούν λύσεις, αποτελεσματικές λύσεις. Και εδώ πρέπει σαφώς και το Προεδρείο να επιληφθεί των προτάσεων αυτό και των σωστών λύσεων. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός αυτών που συμμετέχουν στις ε, διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε τον πολύ υψηλό αριθμό αυτό και εδώ θα πρέπει πραγματικά να τον ε, αμφισβητήσουμε και να ελέγξουμε αν όντως αυτό δικαιολογείται. Είναι πολύ αισιόδοξο ο εισηγητή όσον αφορά το Europal. Και πραγματικά, αν κοιτάξει κανεί τον προπολογισμό, δεν ξέρω αν όλα δικαιολογούνται. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Υπάρχει κάποιος άλλο που θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Γκάιερ. Αγαπητή Ίγγε, το θέμα της ε, κομματικής τοποθέτησης είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε προσεκτικά. Αν οι χριστιανοδημοκράτες θέλουν να έχουν λογικές ε, θέσεις σε αυτά τα θέματα, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το αποδέχομαι, αλλά δεν μπορούμε να δεχόμαστε μια κομματική αντιμετώπιση. Για τα 60.000 ευρώ που αναφέρθηκες, τα οποία δόθηκαν για το σχέδιο αυτό στη Βουλγαρία, εδώ πρόκειται για μια επιδότηση προς την ε, σύζυγο του κυρίου Στάνιτς, του επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βουλγαρίας. Θα μπορούσε κανείς να ελπίσει ότι δεν υπάρχει ε, κάποιος ε, ότι να πιστέψει κανείς ότι αυτό ήταν μια σοσιαλιστική απόφαση, αλλά δεν υπήρχε κανένας ο οποίος ανήκε στο σοσιαλιστικό κόμμα στην ε, δίκηση του Κοινοβουλίου που ενέκρινε αυτή τη δαπάνη. Πώς θα μπορούσε να το ξέρει αυτό όμως η δίκηση του Κοινοβουλίου όταν δεν ήταν ακόμα νυμφευμένη με τον κύριο Στάνιτς η κυρία αυτή που πήρε την επιδότηση. Πώς μπορεί κανείς να αξιολογήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κίνδυνο. Λοιπόν, δεν υπάρχει επομένως η δυνατότητα να καταλήγει κανείς σε τέτοιου είδους ε, συμπεράσματα και δεν είναι σωστό να γίνεται θέμα μια τέτοια περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάια. Κύριε Γκρέσλε έχετε πάλι το λόγο. Μια προσοχή λοιπόν διότι βρισκόμαστε σε ένα είδος εργοταξίου εδώ. Η κυρία Στάνιτσεφ είχε μια επιχείρηση και αν έκανε κανείς ένα κλικ στο ίντερνετ θα έβλεπε ότι αυτή η επιχείρηση, το Active Group, ήταν μεπλεγμένη σε μια υπόθεση διαφθοράς στην Αυστρία. Είχε δοθεί εντολή σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων να καλοποίησει κατά κάποιο τρόπο την εικόνα της ε, Βουλγαρίας προς τον έξω κόσμο και δόθηκε αυτή η εργολαβία κατά κάποιο τρόπο στην μετέπειτα κυρία Στάνιτσεφ. Λοιπόν, οι σχέσεις αυτές που υπήρχαν μεταξύ των εμπλεκομένων θα μπορούσε κανείς να το καταλάβει απλώς με μια σύντομη επισκόπηση στο ίντερνετ. Λυπάμαι λοιπόν κύριε Γκάιερ. Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι ότι έχουν πάρα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε και στην ε, Βουλγαρία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν ένας καθηγητής στην Γερμανία είχε πάρει 80.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ για να παρουσιάσει ε, θετικά κάποιον υποψήφιο ή κάποια ομάδα στη Γερμανία θα είχε γίνει χαμός. Λοιπόν, αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αποδεχτούμε στην περίπτωση της Βουλγαρίας. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι δεν υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Και ο κύριος Στάνισεφ ενδιάμεσα ήτανε ε, έγινε πρωθυπουργό και τώρα είναι μάλλον ο επικρατέστορης υποψήφιος για, για να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Βουλγαρία. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι δεκτά. Είναι για μένα απόλυτα απαράδεκτα και εμένα με ενοχλεί ότι κάποιος προσπαθεί να με πείσει ότι εδώ έγιναν όλα με το σωστό τρόπο. Τα ποσά αυτά λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα να τα, να τα παραγνωρίσουμε και γι' αυτό διαφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κ. Γκάι προηγουμένως. Yeah. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν βλέπω κάποιος να ζητά το λόγο, οπότε θα επιστρέψω τον λόγο στον εισηγητή. Ιβάν. Θα επιθυμούσα να αναφερθώ εν συντομία σε αυτό το σκάνδαλο διαφθοράς, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Διότι δεν αποτελεί αντικείμενο της εκθεσής μου. Σε τελική ανάλυση δεν είμαστε δικαστήριο εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι αφού κυκλοφόρησε το θέμα αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα μέσα, ουσιαστικά εμφανίστηκε ένα άρθρο σε μια ιστοσελίδα και το αντέγραψαν διάφορες άλλες ιστοσελίδες, άλλες εφημερίδες και αυτό που έπρεπε να αποτελήσει αντικείμενο εξέταση σε δικαστήρια μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο σκάνδαλο στον τύπο, πολιτικό σκάνδαλο. Γνωρίζουμε όλες αυτές τις πρακτικές ε, που λαμβάνουν χώρο όχι μόνο στην Βουλγαρία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό η δημιουργία ενό τεχνητού σκανδάλου στον τύπο, με υπερβολές πολιτικές, ε, με αναγωγή του θέματος ευρωπαϊκή κλίμακα. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου όλη η οικογένεια, οι περιβάλλοντες ε, γνωστοί γη, οι κόρε, όλοι βρίσκονται μπλεγμένοι μέσα σε ένα σκάνδαλο διαφθορά. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την επιτροπή πρέπει να τηρούμε τον νόμο και τι διαδικασίε που έχουν θεσπιστεί και πρέπει πάση θυσία να αποφεύγουμε διενέξει ε, πολιτικέ ε, γεμάτης λαϊκισμό τέτοιου είδου. ειδικότερα δύο μήνες πριν από τι εκλογέ. αν είναι να μεταμορφώσουμε τεχνικές εκθέσεις σε πολιτικές ε, οι συζητήσεις θα διαστρεβλωθούν, δεν θα έχουν πλέον νόημα. Ευχαριστώ. Dank. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρέσλε και πάλι. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, πρόκειται για χρήματα το φορολογούμενο. Για κάποιους σοσιαλιστές δεν πρόκειται καν για χρήματα. Αλλά είναι πολιτικό αν θέλει το θέμα. Εδώ πρόκειται παρόλα αυτά για θέμα το οποίο θα έπρεπε να είχε επιληφθεί η δίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κάτι που θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις για το πόθεν έσχες. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να γίνει μία μελέτη, μία ανάλυση και αυτά τα χρήματα, είτε πρόκειται για 60.000 ευρώ, είτε για περισσότερα, είτε για λιγότερα, πρόκειται για ένα ποσό. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει μία ε, ανάλυση του κινδύνου πριν δοθούν αυτά τα χρήματα. Και δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Από τη μία δηλαδή να στηρίζουμε κάποιες πολιτικές ομάδες με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα δώσω τώρα ονόματα. Ο κύριος Γκάιερ ξέρει πάρα πολύ καλά για ποιες πολιτικές ομάδες, σε ποιες πολιτικές ομάδες αναφέρομαι. Εγώ θα υποβάλω την τροπολογία μου, αλλά πραγματικά Ίσως αρχικά η υποστήριξη αυτή να είχε καλό σκοπό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση, η οποία μάλιστα να αναγράφεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για μία ανάλυση κινδύνου πριν δοθούν αυτά τα ποσά. Και θα πρέπει να τηρούνται και κάποια μεγέθη. Λοιπόν, το θέμα εδώ της βουλγαρικής αυτής υπόθεσης, που δεν είναι εξάλλου και η μοναδική, μας δείχνει ακριβώς ότι υπάρχουν αδυναμίες, ότι υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν τέτοιου είδους ε, να προκύψουν και άλλες τέτοιου είδους υποθέσεις. Και θα ζητήσω ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Βλέπω ότι συνεχίζει βημερός αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εδώ βεβαίως το θέμα των πολιτικών παρατάξεων είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο συνολικά το θέμα αυτό για τον οποιονδήποτε Ευρωπαίο φορολογούμενο από τη στιγμή που κάποια χρήματα δεν χρησιμοποιούνται με τον σωστό τρόπο, δεν έχουν το αποτέλεσμα για το οποίο αρχικά είχαν προβλεφθεί, είναι κάτι που σαφώς ε, πλήττει την αξιοπιστία των ε, οργανισμών μας και είναι δική μας υποχρέωση ενώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Διοίκησης να ελέγξει ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο αρχικά είχαν προβλεφθεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και είναι και θέμα, όπως είπατε, αξιοπιστίας. Δηλαδή είναι θέμα του κατά πόσον ο έλεγχος των δαπανών γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο κινητοποιούμε κάποια κονδύλια για να έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σαν Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σίγουρα ε, δεν θα πρέπει να αφήσουμε να γίνει θέμα πολιτικών κομμάτων αυτό το θέμα του ελέγχου των δαπανών. Χρειαζόμαστε έναν αποτελεσματικό έλεγχο και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, εάν θέλει, για να με το θέμα αυτό. Concluzia este cea pe a spus și dumneavoastră, că... Το συμπέρασμα μόλις το είπατε εσείς ο ίδιος, ε, κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται μια τεχνική έκθεση. Πρέπει να βασιστούμε στις ε, διαδικασίες, ε, στα τεχνικά ζητήματα, στους κανόνες που εμείς οι ίδιοι έχουμε υιοθετήσει, οικονομικούς, διαδικαστικούς ε, κανόνες. Δεν πρέπει να πέσουμε στον πειρασμό της προεκλογικής εκστρατείας ακριβώς πριν από τις εκλογές. Καταλαβαίνω τις προθέσεις της κυρίας Γκρέσλε, αλλά θα εμπιστευτώ περισσότερο την άποψη της Γενικής Γραμματείας που δήλωσε ότι όσον αφορά την υπόθεση αυτή για την οποία συζητήσαμε σήμερα δεν υπήρξε πραγματικά σύγκρουση συμφερόντων και από νομική άποψη δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την λογοσύμβαση. Σας ευχαριστώ έντελη για την συζήτηση που είχαμε. Αναμένω τις τροπολογίες με προθεσμία 25 Φεβρουαρίου. Το Μάρτιο θα συναντηθούμε με τους Κιώδης στο Στρασβούργο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε με το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης και περνάμε στο 20. Πρόκειται για τους διάφορους αποκεντρωμένους ε, φορείς. Κύριος Πέτρη είναι εισηγητής. Έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω επίση το Ελληνικό Συνέδριο και τους ε, οργανισμούς για την εξαιρετική τους ε, συνεργασία και συμβούλη. Η απαλλαγή του 2012 για, τις για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς ε, δεν ε, διαφέρει σε κάτι από τα προηγούμενα χρόνια. Όπως θα δείτε στην οριζόντια εκθέση μου για την υλοποίηση του προπολογισμού των οργανισμών για το 2012, πράγματι απομένουν να γίνουν πολλά. Και πάλι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανεπαρκή δημοσιονομικό προγραμματισμό, υπερβολικές μεταφορές ανεπαρκή διαφάνεια, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και τέλος ε, ακατάλληλες επαληθεύσεις χορηγήσεων για να μην πω ότι έλειπαν ουσιαστικά τέτοιες επαληθεύσεις χορηγήσεων. Πρέπει να ενισχύσουμε ουσιαστικά την εκ προτέρων και εκ των επαλήθευση και ειδικότερα την εκ των υστέρων επαλήθευση γεγονός που μας εκπλήσει αρκετά. Προτείνω επίσης τον συντονισμό μεταξύ ορισμένων οργανισμών, ειδικότερα όσον αφορά αποφάσεις ε, που έχουν επιπτώσεις ε, στο πεδίο δράσης ενός άλλου οργανισμού. Αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι μια τέτοια προσπάθεια θα μπορέσει να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ε, με συμφωνία μεταξύ των ίδιων οργανισμών. Δεδομένων αυτών, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους διαφορετικούς ρόλους, λειτουργίες και τους πόρους των διαφόρων οργανισμών και στο γεγονό ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες απαλλαγής. Τι εννοώ με αυτό. Θα το καταλάβετε, θα αναφερθώ σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό τον οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω, να επισημάνω ως θέμα. Ορισμένε φορέ οι καθημερινέ απαιτήσει προ οργανισμού αυτού δεν συνάδουν με την παραδοσιακή διαδικασία απαλλαγή. Και σε ορισμένε περιπτώσει το πολύ περιορισμένο προσωπικό και οι πολύ περιορισμένοι πόροι δυσχεραίνουν ε, για έναν οργανισμό να πληρεί τις απαιτήσει των ε, οικονομικών ελέγχων. Να σε επισημάνω κάποιες περιπτώσεις ε, Πρώτα απ' όλα, ο Οργανισμό των ε, Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τι Ελεκτρονικέ Επικοινωνίε, BEREC, όπω την γνωρίζουμε, να σα το πω σαφώ και ευθέω. Είμαι υπέρ τη αναστολή τη απαλλαγή για την BEREC Τίποτα δεν θεωρείται ότι αποτελεί το αντικείμενο ασφαλμένο πρακτικών οι παραμέλειες, αλλά γενικά οι επιδόσεις της ΜΠΕΡΕΚ το 2012 είναι αρκετά ανεπαρχείς και αυτό με οδηγεί στο να προτείνω κάποια τέτοια οδό. Αν δείτε το σχέδιο εκθεσής μου θα αντιληφθείτε ότι ουσιαστικά κάθε επικεφαλίδα συγγνώμη, σε κάθε περίπτωση τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά το 2012. Η αξιοπιστία των λογαριασμών δεν επαληθεύτηκε. Η νομιμότητα και η διαφάνεια των συναλλαγών, υπέρχουν παρατυπίες. Όσον αφορά τη δημοσιονομική και την οικονομική διαχείριση, μεταφορές, οι δημόσιες συμβάσεις, οι προσλήψεις Πολλά είναι τα θέματα. Και τέλος, ο εσωτερικός οικονομικό έλεγχος. Δεδομένων λοιπόν αυτών, ε, θεωρώ ότι αναβολή είναι ουσιαστικά μια απαραίτητη απόφαση ώστε να δώσει στον οργανισμό χρόνο να πείσει το κοινοβούλιο αυτό ότι μπορεί να διορθώσει τα πεπραγμένα του ότι δεν υπήρχε λόγος να πιστεύουμε εμείς δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι θα ξαναδούμε ποτέ ενό τέτοιου είδου έκθεση από την ΠΕΡΕΚ. Και πραγματικά να σας πω, εδώ μιλάμε για έναν οργανισμό που ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους. Κάθε χρόνο έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα μέσο όρο, ένα... ποτέ δεν είναι τέλειο οργανισμό, αλλά πάντα υπάρχει ένα μέσο όρο. Αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάτι ξεχωριστό. Υπάρχει και ένας άλλος οργανισμός, η Frontex. Έχουμε αυτή τη γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά την ομότητα και την ε, καθαρότητα των συναλλαγών και το ελεκτικό συνέδριο δεν μπόρεσε να εκφράσει άποψη γι' αυτό διότι θεώρησε ότι δεν είχε αρκετά αποδεικτικά στοιχεία και σε ορισμένε περιπτώσει καθόλου προφορίες. Έτσι λοιπόν στην γνωμοδότηση του ελεκτρικού συνεδρίου για παράδειγμα, δεν υπήρχαν επαληθεύσει ε, εξάντε ή εξπόστε εκ των προτέρων ε, εκ των υστέρων για τις ε, συναλλαγές του 2012. Ωστόσο, η ίδια Frontex θεωρεί ότι υπήρχαν επαληθεύσει εκ των προτέρων υπό τη μορφή δηλώσεων που έγιναν από του εθνικού συνοριοφύλακε, τις εθνικές συνοριοφύλακες, αρχέ αρχές και από του ελέγχου που πραγματοποιεί ο ίδιο οργανισμό. Αυτή λοιπόν ε, η αντιπαράθεση στην ερμηνεία οδηγεί σε δύο διαφορετικές απόψει. Κάνω λοιπόν έκκληση προς το ελεκτικό συνέδριο και τον οργανισμό να μας δώσουν μια αμοιβαία αποδεκτή λύση που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα παραδοσιακά κριτήρια οικονομικού ελέγχου καθώς και τις συγκεκριμένες συνθήκες, τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τι οποίε καλείται να δράσει ο οργανισμός αυτός. Αυτό αναφέρω στην οριζόντια έκθεσή μου και αυτό εννοώ όταν αναφέρομαι σε διαφορετικά κριτήρια και διαφορετικά περιβάλλοντα ε, στα οποία δρούν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί. Οι ελλείψεις ε, στους τομείς των προσλήψεων και των εσωτερικών ελέγχων διορθώθηκαν από τη Frontex ίδια πέρυσι. Λαμβάνονται δηλαδή εδώ υπόψη οι πολύ διαφορετικές ε, απαιτήσεις ε, δράσης και οι έλεγχοι που έκαναν οι ίδιοι διόρθωσαν τα πράγματα, ορισμένα από αυτά τα πράγματα το 2013 σύμφωνα και με τις επιθυμίες του ελεκτικού συνεδρίου. Δεδομένων αυτών λοιπόν θα πρότεινα να εκχωρήσουμε την απαλλαγή για τη Frontex. Και τέλος, εν συντομία, Υπάρχει ένας τρίτος οργανισμός που θα ήθελα να αναφέρω πιο συγκεκριμένα, τον EIT για την τεχνολογία πληροφορικής. Υπάρχει και βάση για ε, γνωμοδότηση από το ελεκτικό συνέδριο όσον αφορά την νομιμότητα των ανδράσεών τους και εκεί λείπει η διαφάνεια όσον αφορά τις συναλλαγές του 2010 και του 2011. Πρόκειται για θέματα που ακόμα αποτελούν εφιάλτες για μας. Η εσωτερική έλεγχη σίγουρα δεν ήταν επαρκές. Έλειπαν ποσοτικοποιημένοι στόχοι. Και αυτό θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσέχουμε τι αποτελέσματα επιτυγχάνουμε με τα χρήματα των φορολογουμένων. Πρέπει να γνωρίζουμε τι εννοούμε όταν λέμε αποτελέσματα. Όταν οι στόχοι δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα ποσά, όπως στην περίπτωση του EIT, όταν δεν είναι ποσοτικοποιημένη δηλαδή αυτή η στοχή, είναι δύσκολο να καταλάβουμε αν τα χρήματα που επενδύσαμε απέδωσαν. Αυτό ισχύει για όλους τους οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Στούτο Ανατομίας και Τεχνολογία του, EIT, ε, εμφανιστήκε στην ακρόαση με πια αρκετά πιστικά επιχειρήματα. Εγώ θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να υποβάλουν τροπολογίες, ε, συγγνώμη τα μέλη εδώ, ε, θα μπορούν να, τις επιτροπές θα μπορέσουν να στείλουν μέχρι σε μία εβδομάδα τα σχόλιά τους για την απαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάμαρμε οι αποκεντρωμένοι φορείς πέρσι ήταν στο επίκεντρο του πολιτικού μας ενδιαφέροντος στη διαδικασία της απαλλαγής, αλλά εφέτος δεν είναι τόσο αμφιλεγόμενες, παραμένουν φυσικά σημαντικές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Ναι, ναι, όχι, δύο άτομα. Ο κύριος, De Jong, ο κύριος Μίλτορ και ο κύριος De Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις παρατήρησεις του αν κατάλαβα καλά, τρεις από τους αποκεντρωμένους αυτούς φορείς κινδυνεύουν να μην λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Είναι πάντα χρήσιμο όμως να ακούσει κανείς και την άλλη πλευρά του επιχειρήματος. Παραδείγματος χάρη, σε ό,τι αφορά την Μπέρεκ και τις σοβαρές αυτές κατηγορίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το τι γίνεται σε αυτόν τον φορέα και ποια είναι η τωρινή κατάσταση των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Ο Ντε Ιόγκ. κύριος Ντε Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Πιστεύω ότι όταν είχαμε κάνει την ακρόαση του, της Γενικής Γραμματέως της κυρίας Ντέι από την Κομισιόν μας είχε πει ότι οι φορείς αυτοί είναι ανεξάρτητοι και το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι, που μπορεί να κάνει η Κομισιόν μάλλον, να τους δώσει συμβουλές για το πώς να αποφύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. Αλλά αυτές οι κατευθυντές γραμμές θα πρέπει να εφαρμοστούν βάσει της απόφασης των ίδιων αυτών των αποκεντρωμένων φορέων που μπορούν να διαλέξουν να τις εφαρμόσουν ή όχι. Νομίζω ότι το μόνο θεσμικό όργανο που μπορεί να συζητήσει σε βάθος την κατάσταση των αποκεντρωμένων φορέων είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ με ικανοποίηση βλέπω στην έκθεση του, του εισηγητή ότι το σύστημα ε, παροχή στοιχείων από τις αποκεντρωμένους φορείς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρήζει βελτιώσεων. Είναι πολύ σημαντική αυτή λοιπόν η σύσταση που διατυπώνεται, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω και να εξηγήσει με ποιο τρόπο ακριβώς θα πρέπει να γίνει αυτή η βελτίωση και όχι μονάχα για τους αποκεντρωμένους φορείς αλλά και για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως ο εισηγητής λοιπόν μπορεί να μας, δώσει κάτι περισσότερο ή αλλιώ να υπάρχει ένα τμήμα στην έκθεσή του για τη θέση της Κομισιόν, τη θέση του Κοινοβουλίου και γενικότερα τα θέματα διακυβέρνησης και ευκυβερνησίας των φορέων. Σε ό,τι αφορά την παροχή εκθέσεων Πιστεύω ότι και το ελεκτικό συνέδριο έχει την ίδια εντύπωση όπως και εμείς ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών των αποκεντρωμένων φορέων, δηλαδή ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης τους και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε <clears throat> να κάνουμε μια διαφοροποίηση και να μην κοιτάξουμε να την αποτελεσματικότητα πώς την αντιμετωπίσουμε εμείς, αλλά να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η φορείς είναι πραγματικά μακριά από την κοινή γνώμη. Είναι πολύ σπάνιο και πολύ απίθανο να γίνουν διαδηλώσεις ενώπιον των ε, αποκεντρωμένων φορέων από τους πολίτες γιατί δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν αυτοί οι φορείς. Είναι ένα θέμα λοιπόν λογοδοσίες των αποκεντρωμένων αυτών φορέων σε σχέση με το ευρύ κοινό και αυτό πρέπει να είναι στοιχείο λοιπόν της έκθεσης. Τέλος, σε σχέση με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ανέφερε ο εισηγητής για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, αναφέρονται πολλά στην έκθεση, <clears throat> αλλά βλέπουμε και στα αποτελέσματα να προκύπτουν διαφορετικές ενέργειες λόγω συγκρούσεως συμφερόντων και εδώ δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο οι αποκεντρωμένοι φορείς μπορούν να επαληθεύσουν την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιούν για να καταρτήσουν ε, εκθέσεις. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι σε ό,τι αφορά την ε, υπηρεσία φαρμάκων οι οργανώσεις των ασθενών που χρησιμοποιούνται για τις δοκίμες στα φάρμακα συνδέονται πολλές φορές με φαρμακευτικές εταιρείες. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό επίσης για τη CIPOL Αναφέρεται εδώ στην έκθεση ότι το, το Συμβούλιο θέλησε η ΣΥΠΟΛ να μην είναι στη Χάγη κοντά στη Γεροπόλ αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών ακόμα και αν υπάρχει μια πλειοψηφία της ΛΥΜΠΕ που υποστηρίζει κάτι τέτοιο θα πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε και αυτή τη μάχη και τι θα αποκομίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους ε, εκπροσώπους των αποκεντρωμένων φορέων να σχολιάσουν αυτά τα οποία έχει πει ο εισηγητής. Έχουμε εκπροσώπους της Frontex, IT, BEREC και EFSA που είναι παρόντες. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κατά πόσο κάποιοι από τους εκπροσώπους των αποκεντρωμένων φορέων θα ήθελαν να λάβουν το λόγο. Ποιος θα ήθελα να ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Είμαι από το γραφείο της Μπέρεκ, από την ε, υπηρεσία αυτή. Σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Κομισιόν για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει ότι υπήρξαν ελλείψεις και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην ε, διακυβέρνηση της Μπέρεκ αλλά υπενθυμίζουμε ότι είναι πολύ καινοφανή αυτή η οργάνωση, η ΠΕΡΕΚ. Μόνο το 2011 είναι αυτόνομος φορέας και το 2012 ήταν στη φάση κίνησης και έπρεπε να περατώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Παρά τα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη χρήση των ε, κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα στοιχεία των ετησίων λογαριασμών του 2012 είναι απόλυτα ε, όπως θα έπρεπε να είναι. Η Κομισιόν παρακολουθεί πλήρως το θέμα αυτό και ελέγχει μέσω της Επιτροπής Διοίκησης το ότι η Μπέρεκ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα και έχει αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης με τις κατάλληλες διαδικασίες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου και να λειτουργήσει πιο θετικά. Η πρόταση που έχει γίνει από το γραφείο της Μπέρεκ στο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις αιτήσει του ελεκτικού συνεδρίου έχει συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή όπου συμμετέχει η Κομισιόν. Από τον Ιανουάριο του 2013 το γραφείο της Μπέρεκ έχει συνεργαστεί με την Διοικητική Επιτροπή και έχει δημιουργηθεί μια ειδική μονάδα η οποία θα παρακολουθήσει από κοντά τις απαραίτητες δράσεις για να αντιμετωπιστούν όλα τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν είναι βέβαιη ότι τα μέτρα που έχει υιοθετήσει αυτή τη στιγμή το γραφείο της Μπέρεκ θα επιτρέψει την Μπέρεκ να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι η Μπέρεκ έτσι θα μπορέσει να διαδραματίσει ακόμα σημαντικότερο ρόλο στην υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαίσιου για τις τηλεπικοινωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος να προσθέσει κάτι και για τους άλλους οργανισμούς. Μπορείτε να Σχολιάστε, αν θέλετε οποιαδήποτε από τα ζητήματα που θέτει ο κύριος Σίγητης. Ναι, καλημέρα. Είμαι η Μαρτίν Ρέρα Ρωσινιόλ, προέρχομαι από την Γενική Διεθνή ΕΡΚ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω για τον ε, EIT, τον Ευρωπα... το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Να σας πω ότι η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου περιορίζεται στις δραστηριότητες του 2010 και όχι του 2011. Η Επιτροπή φυσικά αναγνωρίζει τη γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τις δραστηριότητες του EIT που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, αλλά ταυτόχρονα η επιφυλακτική κομισιόν όσον αφορά την πλησίωση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου αυτού. Τι θα ήθελα να απαντήσω λοιπόν ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από τον EIT επικεντρώνονται Πρώτα απ' όλα στη βελτίωση των προτέρων ελέγχων, θέμα που τέθηκε από το Ελληνικό Συνέδριο. Ο ΙΑΙΤ επίση έχει υλοποιήσει μια ε, στρατηγική ελέγχων εκ των υστέρων που μελετήσαμε και επίσης ε, όσον αφορά τις επιδόσεις ε, ο το ΙΑΙΤ μαζί με το ΚΙΚΣ... μιλάμε εδώ για τις χορηγίες ε, για συγκεκριμένους οργανισμούς. Έχει αναπτύξει λοιπόν ένα σύνολο δικτών επιδόσεων Key Performance Indicators, δείκτες ε, κλειδιά. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία έχει τηρήσει του προσανατολισμού που εξέδωσε το Ελληνικό Συνέδριο όσον αφορά τι αδυναμίε του και υλοποίησε ένα σύστημα εσωτερικών ελέγχων και στρατηγικών ελέγχου. Φυσικά η Επιτροπή θα επιτηρήσει την αποτελεσματική υλοποίηση όλων των παραπάνω. Ευχαριστώ. Thank you very much. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ναι, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, ξέχασα να πω ότι όλες οι συντολές ε, ανάκτησης ε, έχουν ενεργοποιηθεί και ανακτηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιο άλλος από κάποιον οργανισμό δεν βλέπω πολύ καλά, ε, που δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Άνευ μικροφόνου. Καλημέρα από ένα Μπύρα από... για το θέμα της Frontex. Το θέμα των ελεγχών εξάντα και εξπόστ συζητείται συχνά σε διοικητικό επίπεδο και η Επιτροπή γνωρίζει τα προβλήματα. Η Κομισιόν χαιρετίζει τις προσπάθειες ε, που έκανε η Frontex για ελέγχους εξάντα και εξπόστ και ειδικότερα την αναθεώρηση της σχετικής πολιτικής από την 1η Ιουλίου του 2013. Έκτοτε έλαβαν χώρα ανεπίσημες επαφές μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης και της Frontex επί του θέματος. Γνωρίζουμε ότι η Frontex έχει ξεκινήσει εκστρατεία ελέγχου ex post το, φθηνό το 2013 που καλύπτει τις δαπάνες και το 2012. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα των οικονομικών ελέγχων είναι πολύ ικανοποιητικά με πολύ χαμηλό επίπεδο σφάλματα. Η διαβίβαση των αποτελεσμάτων στην Γενική Διεύθυνση Home θα λάβει η χώρα στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Η DG Home είναι σίγουρη ότι η Frontex έχει ενισχύσει τις επαληθεύσεις στο μέσο ελέγχων εξ στο στον τομέα των χωριών. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλους τους οργανισμούς. Παρέβλεψα κάποιον. Η κυρία Γκρέσλε και με τον κύριο Σάβαρμε. Ελπίζω ότι δεν μας παρακολουθούν οι εκλογείς μας. αρνούνται τα προβλήματα οι εκπρόσωποι και όπου δεν αρνούνται τα προβλήματα ουσιαστικά τα παρακάμπτουν. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τι πρέπει να κάνουμε για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και για την ΠΕΡΑΚ, γιατί υπάρχουν προβλήματα για το ΕΙΤΕ εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε να γίνονται τα πράγματα χωρίς να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα. Μην περιμένετε ότι του χρόνου θα είναι πάλι εύκολα τα πράγματα. Του χρόνου θα πρέπει να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτα αυτά, ότι δεν είναι εξηγήσει αυτές που μας έχετε δώσει. Όλα αυτά δεν ευνοούν την εικόνα της Ευρώπης. Ο κύριος Σαβαρμέ έχει το λόγο. Σάρβαμα. Ναι, πρόεδρε. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση για τα θέματα αυτά. Γιατί αν διεξέλθουμε το θέμα αυτό σε πέντε λεπτά δεν έχει κανένα νόημα και δεν συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε. Από τη στιγμή που έχουμε αυτή την ευκαιρία θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από την ε, ε, απάντηση της Κομισιόν που εκπροσωπεί την Μπέρεκ. Και επειδή έχουμε τον κύριο Ρέχεμοα, ο οποίος είναι ο διοικητικός διευθυντής, ελπίζω ότι θα είναι σε θέση να συμμετάσχει σε μια πραγματική συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Αλλιώς παίζουμε ένα θέατρο, θέατρο μαριονετών που δεν έχει πολύ νόημα. Νομίζω ότι μας πληρώνουν για να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ας κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και ας έχουμε μια πλήρη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Αν μπορώ να προτείνω κάτι τέτοιο, να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για κάτι τέτοιο. Από τη δική μου άποψη δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο βέβαια. Ακούσατε τις απαντήσεις των εκπροσώπων της Κομισιόν και των αποκεντρωμένων φορέων Ίσως θα έπρεπε να τους απευθύνετε κατευθείαν τα ερωτήματά σας στους αποκεντρωμένους φορείς. Έχουμε επαρκή χρόνο για να το κάνουμε αυτό. Παρακαλώ. Πολύ ωραία κύριε Πρόεδρε. Για την Μπέρεκ. Το βασικό στοιχείο της απάντησής σας ήταν ότι ο φορέας αυτός ήταν μονάχα στη φάση κίνησης το 2012. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και το έχω εξετάσει κάπως ενδελεχώς το θέμα αυτό, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Μπέρεκ ήδη πέρσι και αυτό φάνηκε και στη διαδικασία απαλλαγής της ο κύριος Κέρμπραντ δεν ήταν παρόν εδώ. Ήδη πέρσι υπενθυμίστηκε στην Μπέρεκ ότι υπήρχε ένα πρόβλημα και δεν έχει πράξει τίποτα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ακόμα χειρότερα έχουν γίνει τα πράγματα από την προηγούμενη διαδικασία απαλλαγή. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να ξέρω, είτε από την Γενική Διεύθυνση Connect, είτε από το Διευθυντή του Φορέα, είναι τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το χρόνο, τι έκανε η Μπερακ για να αντιμετωπίσει αυτές τις κριτικές. Παρακαλώ. Λέγομαι Ρέιν Φαντέι από την GD Budget. Πιστεύω ότι μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες και μπορούμε να δώσουμε και στους φορείς αυτούς τους ίδιους αλλά και στη Γενική Διεύθυνση να εξηγήσουν και να απαντήσουν δίνοντας πολύ συγκεκριμένες και ισορροπημένες ε, απαντήσεις στις ερωτήσεις της Επιτροπής σας. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να είσαστε έτοιμοι για την υποβολή τροπολογιών, να σας υποβάλουμε όλες αυτές τις απαντήσεις. Ναι, λέει ο πρόεδρος, αλλά βρίσκομαι σε μία λίγο περίεργη στάση. Θυμάστε την έκθεση Μακοβέη. Με πολύ επικριτικές ερωτήσεις. Και τότε, μάλιστα, είχαμε πει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λίγο πιο ρεαλιστικό, πιο συγκεκριμένο, όχι τόσο εντυπωσιακό αντιμετώπισης αυτών των ε, θεμάτων. Αλλά θα πρέπει και εσείς να πάρετε λίγο πιο στα σοβαρά την ε, Επιτροπή μας. Εάν δεν θέλετε να μας δίνετε εδώ απαντήσεις, ο εισηγητής ε, υπέβαλε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Το ίδιο και το ελεκτικό συνέδριο. Περιμένουμε λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις από εσάς. Μπορεί να γίνει γραπτά, βεβαίως. Επανερχόμεθα δηλαδή σε μια διαδικασία την οποία θέλαμε να ξεπεράσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πολύ θα ήθελα την επόμενη φορά να χρησιμοποιήσετε την ευκαιρία που σας δίνουμε να είστε εδώ παρόντες, έτσι ώστε να μας δείξετε ότι μας παίρνετε και λίγο στα σοβαρά. Θα ξαναδώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μπορούμε να θέτουμε εδώ συγκεκριμένε ερωτήσει και να παίρνουμε απαντήσεις. Εάν όχι, εάν η Επιτροπή αποφασίζει ότι ε, δεν γίνεται κάτι τέτοιο, να επιλέξουμε μια άλλη διαδικασία. Κυρία Γκρέσλα, κοιτάξτε, είμαστε όλοι εδώ για να μάθουμε κάποια πράγματα. Και εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί μας λέτε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μας δώσετε τις απαντήσεις. Λυπάμαι, λυπάμαι. Δεν μας παίρνετε στα σοβαρά. Και εμείς μπορούμε αυτό να το διαπιστώσουμε και να επιλέξουμε όντω κάτι άλλο, μια άλλη διαδικασία. Είστε εδώ. Γιατί δεν μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Τις ερωτήσεις τις γνωρίζατε. Πραγματικά, θέλω να σας πω ότι έχω αρκετά εκνευριστεί. Πραγματικά, φτάνει, φτάνει. Ε, εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τους ε, ψηφοφόρους μας. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν λίγο. Ελπίζω να μην μας άκουσε και να μην μας είδε κανείς σήμερα εδώ. Είναι κάτι που πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ντότσου. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η κυρία Γκρέσλε. Δεν θέλω να γίνομαι συναισθηματικός. αλλά είμαι ένας ε, νέος ευρωβουλευτής ε, μόλις πέντε ετών εδώ και πέντε χρόνια συμμετέχω στις ε, συζητήσεις που αφορούν τις απαλλαγές άλλοι συναδέλφοι κάνουν την ίδια δουλειά εδώ και πάνω από 15 χρόνια η αίσθηση που έχω εγώ είναι η αίσθηση που είχα όταν βρισκόμουν στο πανεπιστήμιο συγγνώμη, στην ε, Επιτροπή ότι οι οργανισμοί θεωρούν ότι οι ευρωβουλευτές είναι ανόητοι. Και η συζήτηση αυτή λαμβάνει χώρα με τέτοιο τρόπο ουσιαστικά αν σε ένα κράτος μέλος λάμβανε χώρα μια ίδια συζήτηση όλοι οι οργανισμοί, το Συμβούλιο, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο θα έλεγαν στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στι κατοχώρε στην Ουγγαρία πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ενώ ταυτόχρονα βρισκόμαστε εμεί εδώ ως εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και κάνουμε διάλογο μεταξύ κοφών. Τι θέλω να ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Σιγητή. Είναι σημαντικό όταν συζητάμε για τις απαλλαγές ε, Είναι σημαντικό ίσως όλες οι απαλλαγές να, να στάλουν. Θα πρέπει να στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα ότι οι οργανισμοί μπορούν να κάνουν με αυτό που θέλουν αυτοί, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι. Έχουμε καμιά τριανταριά περίπου νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, αλλά μπορεί ενδεχομένω να μου το πούν άλλοι βουλευτές. Υπάρχει τέτοιο πλήθος οργανισμών πρέπει να δούμε κατά πόσο αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι εγώ θα υποβάλω τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. να ανασταλεί η απαλλαγή όλων των οργανισμών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα είναι το αίτημά μου. Όχι μόνο να ανασταλεί η απαλλαγή των οργανισμών που παρουσιάζουν πρόβλημα. Είναι απλά διαδικαστικό το ζήτημα. Υπάρχει ήδη το ιστορικό, διότι για την απαλλαγή του Συμβουλίου έτσι κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν είναι λόγω του περιεχομένου, αλλά λόγω της διαδικασίας. Αναστέλουμε την απαλλαγή για αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τους εκπρόσωπους ε, των φορέων. Θα σας ξαναδώσω το λόγο, ο κύριος Ντεγιόν καταρχήν. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι. Καταρχήν είπα ότι μετά τις παρατηρήσεις της Catherine Days μέσα της Επιτροπής ανησύχησα ότι δηλαδή η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να απαντήσει, είπατε δεν υπάρχει διάλογος αυτό δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί, γιατί το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε και του χρόνου. Νομίζω ότι μετά από τρία χρόνια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε πιο ενεργοποιημένοι και εγώ δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω και να δώσω απαλλαγή εάν δεν έχω όλες τις πληροφορίες που ζητώ. Κύριος Γκάιερ, συμφωνώ και εγώ. Δεν πρέπει να είστε τόσο προκλητικοί με την Επιτροπή μας. Μια φορά το χρόνο συναντώμεθα εδώ μετά από το τέλος της διαδικασίας για την απαλλαγή. Και ουσιαστικά αυτή η διαδικασία έχει σαν σκοπό να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Αν αυτή η διαδικασία που έχει αυτό το σκοπό αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο, με τέτοια στάση από μέρους των ε, αποκεντρωμένων φορέων, νομίζω ότι δικαιολογείται αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς γίνεται η κατανομή καταρχήν των εργασιών μεταξύ Επιτροπής και εκπροσώπων των διαφορών αποκεντρωμένων φορέων. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι παίζεται και ένα παιχνίδι. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ίσως εδώ υπάρχει μια παρανόηση παρόλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τους εκπροσώπους και της Επιτροπής και των φορέων αν μπορούν να δώσουν κάποιες περισσότερο σοβαρές ε, απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Βεβαίως και τα κονδύλια αυτά που αφορούν ουσιαστικά τους αποδροκημένους φορείς είναι αντικείμενο επικρίσεων. Δεν ζητούμε εδώ να υπάρξει μια πλήρης αλλαγή. Υπήρξε πολιτική απόφαση των κρατών μελών όταν ιδρύθηκαν αυτοί οι φορείς είναι ίσως πολλές φορές θέμα χρησιμοποίησης κονδυλίων, είτε κατεύθυνσης, είτε πολιτικής. Αυτό βεβαίως δεν είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ίδιων αυτών των ε, οργανισμών, αλλά σίγουρα είναι στη δική σας αρμοδιότητα να δώσετε ικανοποιητικές απαντήσεις, απαντήσεις που μπορεί να ικανοποιήσουν και εμάς αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν ξέρω ε, Κάποια στιγμή πάντως πρέπει να συντονίσετε τις απαντήσεις σας έτσι ώστε να είναι ικανοποιητικέ και για μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήταν πρόθεση μας να αποφύγουμε κάποιες ερωτήσεις ή να μην ε, δώσουμε απαντήσεις εφόσον ήταν δυνατόν. Αν κατάλαβα όμω τη διαδικασία σωστά, ε, οι οργανισμοί που κλήθηκαν στην προηγούμενη ε, συνεδρίαση, προσκλήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΚΟΝΤ και δεν προσκλήθηκαν σε αυτήν εδώ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η Κομισιόν ήταν εκεί για να απαντήσει. Η Κομισιόν βρίσκεται εδώ για να απαντήσει σε δικό τη επίπεδο τις ε, ερωτήσει, ε, Μπορούμε να παράσουμε γραπτές απαντήσεις ε, ακόμη και τελευταία στιγμή. Για παράδειγμα για την ΠΕΡΕΚ μπορείτε να λάβετε γραπτές απαντήσεις σήμερα. Δεν προσπαθούμε λοιπόν να αποφύγουμε να απαντήσουμε. Απλά προσπαθούμε να δυσφαλίσουμε ότι οι απαντήσεις μας θα είναι πιο πλήρες και πιο ικανοποιητικέ. Θα θέλαμε να προσθέσουμε κάτι για το EIT, οπότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Παρακαλώ. Ναι. Ο διευθυντής του φορέα μας ήρθε στις 20 Ιανουαρίου στη συνεδρία που αναφέρατε και είχε στείλει τις απαντήσεις στα 43 συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία είχατε θέσει. Βέβαια, αν έχετε πρόσθετες ε, ερωτήσεις ή αν αυτές οι απαντήσεις δεν σας ικανοποιούν, είναι προφανές ότι και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και η αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση είναι έτοιμοι να απαντήσουν το ταχύτερο δυνατόν για να μην δοθεί η εντύπωση ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες του φορέα και της Κομισιόν, αλλά αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις πέραν των 43 ερωτήσεων ή θέλετε μια διευκρίνηση για κάποια από αυτές τις 43 ερωτήσεις που έχουν συζητηθεί στις 20 Ιανουαρίου. Είμαστε στην απόλυτη διάθεσή σας. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι περισσότερο νομίζω σήμερα, αλλά θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή εφόσον το επιθυμεί. Ας χαλαρώσουμε λέει ο εισηγητής. Πρώτα απ' όλα εάν ε, γίνουμε υπερβολικοί σε αυτή τη συζήτηση και αρχίσουμε να λέμε ότι όλη η διαδικασία απαλλαγή ε, δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε μπορούμε κάλλιστα να τα μαζέψουμε και να φύγουμε από εδώ. Το πρόβλημα δεν είναι διαδικαστικό τόσο πολύ. Υπάρχουν κάποια σαφή βήματα και το πρόβλημα μου, αυτό που αναφέρω δηλαδή σήμερα, είναι ότι ουσιαστικά πρέπει να κρατήσουμε μια απόσταση και να δούμε τους 31 οργανισμούς ε, από μια απόσταση, μια αλφα απόσταση. Το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται αυτή η άσκηση είναι ότι όταν προσπαθούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο, σε συμφωνώ απόλυτα, πρέπει να αναμένουμε, όπως είπε ο κ. Γκάια, καλύτερο αποτέλεσμα κάθε έτος. Δηλαδή κάθε έτος το αποτέλεσμα πρέπει να βελτιώνεται συνολικά όσον αφορά τις επιδόσεις για παράδειγμα. Οι επιδόσεις των οργανισμών πρέπει να βελτιώνονται ετησίως. Αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξει εν μια νυχτή. Αυτό λοιπόν που προσπαθώ να τονίσω εδώ, να έχουμε μια γενική εικόνα από κάποια απόσταση και να δούμε κατά πόσο ξεχωρίζει κατά κάποιο τρόπο κάποιος οργανισμός ε, και κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους οργανισμούς που ξεχωρίζουν ως υποδείγματα για τους άλλους. Η διαδικασία ακροασής πήγε πολύ καλά και αυτό που δεν καταλαβαίνω εδώ είναι η Κομισιόν, οι οργανισμοί λένε σήμερα στις 18 Φεβρουαρίου ότι καθίστε λίγο, ας ε, πάρουμε άλλη μια εβδομάδα, διότι τα σχέδια έκθεσης, ε, ξέρετε, τυπώθηκαν πριν πολύ καιρό. Όλοι πρόλαβαν να τα διαβάσουν και γνωρίζω ότι ο οργανισμός που ξεχώρισε μεταξύ όλων των υπολείπων, οι οργανισμοί που ξεχώρισαν μετά το, όλων των υπολείπων ξεχώρισαν διότι βασιστήκαμε σε πολύ προσεκτική εξέταση. Κάποιε απαντήσει που έλαβα για το EIT για παράδειγμα με ικανοποιούν. Μετά από την ακρόαση είχαμε το σχέδιο έκθεση. Ε, τυπώθηκε αυτό. Μπορεί να διαβάσει κανεί το σχέδιο έκθεση και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ αυτό που βρίσκω δυσάρεστο όλο ζήτημα είναι η Μπέρεκ. Θα υπάρχει κάποια σημεία κρίσιμη σημασία με το EIT και υπήρχαν και με το EOBA αλλά τελικά επεξηγήθηκαν μια χαρά στην ακρόαση. Όλα λοιπόν είναι... Βγάζει νόημα δηλαδή όλη η υπόθεση. Έχουμε μια γενική εικόνα όπου εξετάζουμε μία, έναν ένα τους οργανισμούς. Στην αρχή υπήρχαν 7 οργανισμοί που δεν μας ανησυχούσαν για τίποτα, οπότε αφήσαμε στο πλάι τις εκθέσεις. Οπότε βήμα, βήμα φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε αυτά τα ζητήματα του 2012. Ε, τα ζητήματα των οργανισμών που δεν είχαν ικανοποιητικές επιδόσεις. Και μάλιστα ακόμα και αφού εξετάσαμε όλους τους οργανισμούς, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έχουμε τα σχέδια εκθέσεων, έχουμε μία εβδομάδα για τις τροπολογίες και γνωρίζουμε ότι αν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η έκβαση για την ΠΕΡΕΚ θα είναι εξαιρετικά δυσχερή. Ε, δεν ξέρω τι να πω για του άλλου οργανισμού, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη και ο εισηγητή έχει μόνο μία ψήφο 18 Μαρτίου, ε, μην το ξεχνάτε αυτό. Ε, μην το παίρνετε λοιπόν ελαφρά την καρδία. Γιατί δεν ξέρετε τι θα βγει από αυτή την Επιτροπή 18 Μαρτίου. Ειλικρινά λοιπόν σας παροτρύνω και ελπίζω να Μα ενημερώσει σχετικά η Μπέρε γιατί μίλησα με τον κύριο Ρέγματ πριν από αυτή τη συνάντηση και ε, είναι έτοιμο να μα πει ποια θα είναι τα βήματα. Με ποιο τρόπο ίσω το ελεκτικό συνέδριο παρανόησε κάτι, αν εγώ παρανόησα κάτι. Η πραγματικότητα δεν είναι... Αν η πραγματικότητα δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του σχεδίου έκθεση, πρέπει να μα το πείτε τώρα, διότι υπάρχει μια προθεσμία την επόμενη Τρίτη και μετά ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Yeah, okay. Uh, now I give the floor. Ξαναδίνω το λόγο στους αποκεντρωμένους φορείς. Η Μπέρεκ θέλει να πει κάτι. Βεβαίως, ελάτε. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το πρακτέο. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα. Θα πρέπει να περιμένουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω να υπάρξει σκάνδαλο θηρία όμως γύρω από τη διαδικασία ε, απαλλαγής λόγω ορισμένων προβλημάτων με τους αποκεντρωμένους φορείς. Δεν θα ήταν σωστό ή αναλογικό. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη μονάχα. Και πρέπει να το δούμε το θέμα ευρύτερα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου ξαναδίνετε το λόγο. Τι να σας προτείνω εγώ και πιστεύω ότι θα αφήσει όλα τα μέρη. Η Κομισιόν θα μελετήσει τα κύρια ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου και θα προσπαθήσει εν συντομία να τα εξηγήσει χωρίς να μπει σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσει λοιπόν για κάθε εύρημα να εξηγήσει τις δράσεις της Μπέρεκ ε, σε συνεργασία με την Διοικητική Επιτροπή μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση ώστε να διευκρινιστούν τα διάφορα ζητήματα. Ελπίζω να συμφωνείτε. Το πρώτο σχόλιο που έθεσε το ελεκτικό συνέδριο ήταν ότι λυπάται που το λογιστικό σύστημα του οργανισμού δεν έχει ακόμα επαληθευτεί. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ε, το λογιστικό σύστημα του γραφείου Μπέρεκ ε, σήμερα έχει επαληθευτεί. Έχει επικυρωθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο έβριμα του ελεκτικού συνεδρίου ήταν ότι το σχόλιο περί της νομιμότητας ε, των συναλλαγών και το ελεκτικό συνεδρίο λυπάται που οι μεταφορές δεσμεύσεων 10% δεν αντιστοιχούσαν στις νόμιμες δεσμεύσεις και υπήρχε θεώρησε, παρατυπία μεταξύ δεσμεύσεων Και έτσι λοιπόν το γραφείο Μπέρεκ ε, ανέφερε τις πληροφορίες σε ένα εγχειρίδιο και σε ένα στη διαδικασία τώρα ακολουθείται από όλους τους αρμόδιους οικονομικούς συντελεστές στο οικονομικό κύκλωμα, στο κλείσιμο του οικονομικού έτους 2013 με ιδιαίτερη εστίαση στη σωστή πρόβλεψη των απαραίτητων μεταφορών και των ορθών νομικών δεσμεύσεων αυτό είναι το δεύτερο έβριμα. Το τρίτο έβριμα του ελεγκτικού συνεδρίου εστιαζόταν στην διαχείριση του προϋπολογισμού και των οικονομικών. Το δικαστήριο σημείωσε ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό του 2012 οδήγησαν σε ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού μόλις 63,4% και δεσμεύσεις πληρωμών και εκτέλεση ήταν 66,16. Η Κομισιόν παρακολουθεί την υλοποίηση του προπολογισμού του 2013 και το 2013 συνεχίστηκε η παρακολούθηση του προπολογισμού από τη Γενική Διεύθυνση και το γραφείο της Μπέρεκ. Αυτή τη στιγμή οριστικοποιούνται οι λογαριασμοί του 2013, οριστικοποιήθηκαν χθε, αν δεν κάνω λάθο. Η υλοποίηση του προπολογισμού ήταν σε ποσοστό βελτιωμένο 89,15% και 76%. Δεν μπορούμε λοιπόν να διορθώσουμε το παρελθόν, αλλά μπορούμε να καταγράψουμε ε, βελτίωση στο ε, έτος 2013. Ειδικότερα όσον αφορά τις μεταφορές και τις αναλήψεις υποχρεώσεων, Ορισμένες αναλήψεις υποχρεώσεων ε, ακυρώθηκαν και λοιπά το ελεκτικό συνέδριο αυτό και επίσης ανέφερε ότι ορισμένα κονδύλια δεν χρησιμοποιήθηκαν και χρειάστηκε, κάποιες πιστώσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν και χρειάστηκε να ακυρωθούν και επίσης ε, η καθυστέρηση μεταφοράς το 2013 ήταν ε, υψηλή 19% του συνόλου. Έτσι λοιπόν πιστεύει ότι το γραφείο Μπέρεκ δυσκολεύεται όσον αφορά στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Όπως εξήγησα, πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς και σαφής ορισμός αρμοδιοτήτων που είχαν συμπεριληφθεί στο σχετικό εγχειρίδιο και έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους οικονομικούς συντελεστές. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στους λογαριασμούς 2013 από αυτή τη στιγμή οριστικοποιούνται οι μεταφόρες των commitment appropriations ε, από το 2013 ήταν 13% ε, του συνόλου, λιγότερο λοιπόν από το 2012. Υπάρχει βελτίωση συνεπώς. Ένα άλλο έβριμα αφορούσε τις ε, ε, δημόσιες ε, συμβάσεις και τις προσλήψεις. Βασίστηκε λοιπόν η Μπερέξ στο οικονομικό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων ε, και ορίζεται ο νέος ρόλος του υπευθύνου προμηθειών που υποστηρίζει την όλη διαδικασία προμηθειών όσον αφορά τις προσλήψεις. Έχει αναπτυχθεί μια διαδικασία υποστήριξης της διαδικασίας και έχει κοινοκοποιηθεί προστήριξη το 2013. Οι ανακοινώσει και θέσεων στον οργανισμό ενημερώθηκαν βάσει των παρατηρήσεων της ΕΚΑ. Όσον αφορά την πολιτική κινητών τηλεφώνων, η πολιτική τηλεπικοινωνιών ε, εισήχθηκε αυτό το σκοπό το 2013 και ενημερώθηκε το 2014. Η πολιτική αυτή ορίζει κανόνες για την παροχή κινητών τηλεφώνων σε μέλη του προσωπικού που τα χρειάζονται για τα ταξίδια τους. Όσον αφορά την πολιτική του Ταμείου, έχει ολοκληρωθεί η σχετική σύμβαση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής σύμφωνα με τον νέο οικονομικό κανονισμό. Όσον αφορά τους εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους, όπου το ελεγκτικό συνέδριο θέτει το ζήτημα ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους. Το γραφείο Μπέρεκ έχει υλοποιήσει το πρότυπο των εσωτερικών ελέγχων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που ορίστηκε μαζί με τις υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου. Το γραφείο Μπέρεκ ε, έκανε προσπάθειες το 2013 σε συνεργασία με διάφορους ε, βοηθούς για να βελτιώσει το πρόγραμμα εργασίας του γραφείου Μπέρεκ ώστε να επισημοποιήσει τη διαδικασία με σαφή βήματα, σαφείς αρμοδιότητες και σαφή χρονοδιαγράμματα. Πολλές διαδικασίες ε, επίσης ορίστηκαν στο εγχειρίδιο λογιστικής και στο οικονομικό εγχειρίδιο κοινοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από όλους τους οικονομικούς συντελεστές. Επιπλέον, η Μπέρεκ στον τομέα των ε, ενημέρωσης και των επικοινωνιών έχει αναπτύξει μια πολιτική ασφάλειας ε, με διάφορε διαδικασίες διαχείρισης. Αυτή είναι μια σύντομη απεικόνηση όλων των δράσεων του γραφείου Μπέρεκ ε, στο τρέχον έτος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο? Από τους αποκεντρωμένους φορείς? Όχι. Νομίζω ότι ήταν πιο ενδελεχής και πλήρης αυτή η παρουσίασή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή, μήπως θέλετε να κάνετε κάποια τελικά σχόλια. Ναι, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω για τις λεπτομεριακές πληροφορίες που δόθηκαν τώρα για τα περισσότερα θέματα που αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης. Από τη δική μου πλευρά λοιπόν δεν έχω να πει τίποτα, απλώς ευχαριστώ όλους τους εμπλεκομένους και θα εξετάσουμε προσεκτικά τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και θα καταλήξει η Επιτροπή μας στην τελική της θέση για την απαλλαγή. Ευχαριστώ. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε και αυτό το σημείο της ημέρησης διάταξης. Θα ήθελα να ζητήσω να λάβει το λόγο κυρία Αγιάλα Σέντερ. Εάν δεν είναι παρούσα, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε το απόγευμα. Α, δεν έχουμε τη συνάντηση το απόγευμα. Ήταν το τελευταίο σημείο. Μα αν δεν είναι εδώ η κυρία Αγιάλα, να προσπαθήσω να την ε, εντοπίσω, λέει η γραμματεία. Α, εδώ είναι η κυρία Αγιάλα. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ έχει το λόγο λοιπόν. Στην έκθεση ΠΙΦ έχετε το λόγο. έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2012 ήταν ένα κομβικό έτος σε σχέση με πρωτοβουλίες που είχαν σαν στόχο να βελτιωθεί ο αγώνας κατά κάθε μορφής ατασταλίας και κυρίως απάτης κατά του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, η Κομισιόν έχει παρουσιάσει μια πρόταση που μας φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για οικονομικά θέματα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η πρόταση, το έχουμε συζητήσει ήδη προηγουμένως και αυτό μπορεί να είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης βελτιώθηκε η κατάσταση με τον νέο κανονισμό της ΟΛΑΦ και για τα θέματα διακυβέρνησης οικονομικής που μπορούν να είναι ένα σημαντικό εργαλείο κατά των απατών και επίσης συγχρόνως υπήρξε η πρόταση της δημιουργίας παράλληλα με την ε, δημιουργία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα υπήρξε η πρόταση για την προστασία των οικονομικών συμφέρων με τη χρήση του ποινικού δικαίου. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες πλαίσιο μέσω του οποίου μπορούμε να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση σε σχέση με την τυπολογία των αδικημάτων σε ελάχιστες κοινέ ποινές, ένα λοιπόν θεμελιώδες πλαίσιο για να έχουμε μια αξιόπιστη αντιμετώπιση των ατασταλιών και των απατών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χάρη λοιπόν στην παρουσίαση αυτή της έκθεσης τη Κομισιόν έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με τα θέματα αυτά, χωρίς ε, αν θέλετε, μεγάλα άλματα και εντυπωσιακές ενέργειες, βλέπουμε ότι υπήρξε μια μείωση σε σχέση με την εντοπιζόμενη απάτη, 30 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά τα κονδύλια ε, αυτά. Είδαμε λοιπόν όμως και σε ό,τι αφορά τις καταβολές πληρωμών να υπάρξει και μια μεγαλύτερη ε, έκταση σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία ε, απατών, αλλά δεν είναι τεράστιο το πόσο αυτό τώρα μας οδηγήσει σε έκτακτες ενέργειες. Μέσα στα πλαίσια αυτής της έκθεσης για τον αγώνα κατά της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμείς παραδοσιακά προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις ε, απάτες στον τομέα των δαπανών. Εδώ είναι τα πράγματα λιγάκι δύσκολα, τα κράτη-μέλη εκτελούν το 80% του προϋπολογισμού, εμείς στη συνέχεια προσπαθούμε μέσω της Κομισιόν να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα εκτελέσουν σωστά τον προϋπολογισμό αυτό ε, στον τομέα των ε, δαπανών, <clears throat> αλλά και στον τομέα των εσόδων, όπου όπως είπα παρουσιάστηκε μια βελτίωση, για να μειωθούν τα σφάλματα και οι ατασταλίες καθώς και οι απάτες. Είναι αλήθεια όμως ότι στον τομέα που υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, είναι ο τομέας της συλλογής εσόδων. Είδαμε ότι μέσα στις διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις πολιετές, πολιετές δημοσιονομικές προοπτικές, εντοπίστηκε με πιο συγκεκριμένο και αυτό τρόπο η κατάσταση αυτή και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ζητούν να κάνουμε κάτι για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή που είναι το τμήμα που έχει να κάνει τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μειώνεται όλων και περισσότερο και γι' αυτό εμείς Κάθε φορά οι προσπάθειές μας για την καταπολέμηση ε, των απατών αφορά ένα όλο και μικρότερο προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις, ε, τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε σαφές από τη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές ότι πρέπει να προβούμε σε ριζικές αλλαγές και αυτό το τόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που πρέπει να ανταποκρίνεται στις ε, επιδιώξεις των πολιτών. Έχουμε λοιπόν έναν κακοήθη όγκο ο οποίος είναι η φοροαπαφυγή και φοροδιαφυγή. <clears throat> Αυτό επηρεάζει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σε επίπεδο 2.000 ευρώ το χρόνο για κάθε πολίτη. 2.000 είναι αυτά τα οποία χάνονται λοιπόν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό όταν σκεφτούμε πόσο μεγάλε είναι οι περικοπές που έχουν γίνει στις δημόσιες προϋπολογισμούς, αποδοχές, συντάξει κτλ. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Επίσης, μέσα στην φοροδιαφυγή πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στην ε, απάτη για το ΦΠΑ. Με τη μεγάλη κρίση που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τις επιπτώσεις για πάρα πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως νότια κράτη, βλέπουμε να υπάρχει σημαντική ε, γκρίζα οικονομία στις χώρες αυτές. Είχαμε στην αρχή καταφέρει να τις συρρυκνώσουμε, αλλά τώρα ερχόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Αναπτύσσονται νέα προβλήματα με τις καθυστερήσεις στην καταβολή ΦΠΑ, με τα σφάλματα που καλύπτουν το 1,5% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ακριβώς που υπόκεινται σε απάτες ΦΠΑ. Και υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των ποσών που εισπράττονται έναντι αυτών που θα έπρεπε να εισπράττουν. 15 δισεκατομμύρια είναι υπό υποψία, αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, και η Ιταλία είναι χώρες όπου υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ του ποσού που πρέπει να εισπράτεται και αυτό που εισπράτεται. Λέει η Κομισιόν ότι δεν είναι μονάχα θέμα απάτης, υπάρχουν οι χρεοκοπίες πάρα πολλών επιχειρήσεων και μικρόμεσων επιχειρήσεων. Υπάρχουν και θέματα νομικών διαμάχων, γιατί ένας τρόπος είναι <clears throat> να αποφεύγει κανείς, υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να αποφύγει κανείς για ένα διάστημα τουλάχιστον την, ε, τον ΦΠΑ και εδώ χρειάζονται αλλαγές στις ε, οδηγίες για τα θέματα αυτά. Υπάρχει και πάλι ένα παράδοξο ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνουν την ικανότητά τους <clears throat> να καταγγείλουν και να διαπιστώσουν ατασταλίες, ακόμα και ατασταλίες που δεν είναι απάτη αλλά είναι ε, σφάλματα και βρίσκουμε λοιπόν σε επίπεδο διαφάνεις. Το πρόβλημα είναι ότι μετά, όταν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η Κομισιόν δεν κάνει τα απαραίτητα για να μπορέσει να ανακτήσει τα ποσά αυτά. Και η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να δει με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί και να βελτιωθεί η κατάσταση από τα κρατη και να μην υπάρξει περαιτέρω απάτη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εντοπιστεί και αυτή η θέληση των κρατών μελών και επίση η Κομισιόν έχει προβεί σε μια περισσότερο σε βάθος ανάλυση σε σχέση με τις ατασταλίες που έχουν ταξινομηθεί ως <clears throat> απατηλές. Δεν είναι λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει μονάχα οι ατασταλίες, αλλά κυρίως αυτές οι ατασταλίες οι οποίες έχουν χαρακτήρα απάτης. Η δική μας πρόταση λοιπόν <clears throat> υποστηρίζει τα νέα αυτά εργαλεία της Κομισιόν. Τονίζουμε το ότι πρέπει να αναγνωριστεί <clears throat> και η προσπάθεια των κρατών μελών που καταβάλουν μια προσπάθεια για να εντοπίσουν καλύτερα τις απάτες. Βλέπουμε ότι σε ορισμένε πιο χτυπητές περιπτώσεις υπάρχει και κάποιο τελικό συμπέρασμα σε σχέση με τη δημοσιονομική περίοδο μέχρι το 2006. Και επειδή έχουμε αιτήσιες <laughs> εκθέσεις, αλλά ένα προϋπολογισμό ο οποίος έχει πολύ χαρακτήρα, Υπάρχουν πολλές ε, διορθώσεις οι οποίες θα πρέπει να επέλθουν. Χωρίς λοιπόν να μπούμε σε όλα αυτά τα θέματα που είναι θέματα απάτηση, υπάρχουν τα σφάλματα, υπάρχουν καθυστερήσεις που συσσωρεύονται στο τέλος κάθε προϋπολογιστικής περίοδου. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούμε να έχουμε μεθόδους οι οποίες καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού η διαδικασία αυτή για τον εντοπισμό των σφαλμάτων να μην οδηγεί σε συσσόρευση διορθώσεων και ανακτήσεων που υπόκειται σε καθυστερήσεις. Πέραν αυτών ζητούμε στην έκθεσή μας, και εγώ το τονίζω ιδιαίτερα, φυσικά εσείς με τις τροπολογίες σας μπορείτε να το βελτιώσετε ακόμα περισσότερο, ζητούμε να υπάρχει μια καλύτερη εφαρμογή των συστάσεων που κάνει η Κομισιόν στις ετήσιες εκθέσεις της και που συνέχεια τα κράτη-μέλη δεν τις εφαρμόζουν πλήρως. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε στα κράτη-μέλη να μας εξηγήσουν καλύτερα, να μας παρουσιάσουν την επιχειρηματολογία τους όταν αποκλίνουν από τις προτάσεις της Κομισιόν. Θέλουμε επίσης η μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ που έγινε στο τέλος του 2011 και στο τέλος του 2012 δεν είχε εφαρμοστεί ακόμα πλήρως Ελπίζουμε ότι η μεταρρύθμιση στο σύστημα ΦΠΑ θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα εφόσον και από τα κράτη-μέλη υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ταχείας αντίδρασης, η απλοποίηση των δηλώσεων ΦΠΑ θα μπορέσουν να αποδώσουν καρπούς. Μας ανησυχεί βέβαια ότι οι τομείς όπου εξακολουθούν να υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ατασταλίες και σε απάτες είναι τομείς όπως είναι η γεωργία, παραδείγματος χάρη, ενώ στη γεωργία ήδη είχαμε αναφέρει όταν συζητήσαμε για τα θέματα της μετάβασης από τον πρώτο, πυλώνα στο δεύτερο, είχαμε πει ότι εκεί που υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος στα θέματα αγροτικής ανάπτυξης εκεί πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις άμεσες πληρωμές όπου υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για να αποτρέψει κανείς την απάτη. Επίσης και στον τομέα συνοχής έχουν διαπιστωθεί προβλήματα παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι με την τωρινή νομοθεσία η οποία έχει θεσπιστεί με τους νέους κανονισμούς και με την συρρήκνωση των προθεσμιών θα μπορέσει να εντοπίσει καλύτερα την απάτη. Επίσης, σε ό,τι αφορά την προεταξιακή χρηματοδότηση, μας λέει η Κομισιόν ότι εφόσον καταρχήν μερικά κράτη έχουν γίνει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παίρνουν πλέον προενταξιακή βοήθεια και υπήρξε μια θετική πορεία απόκτησης γνώσεων σε σχέση με τη λειτουργία αυτών των προταξιακών χρηματοδοτήσεων. Για τις διεθνείς συμφωνίες ζητάμε πάντα να υπάρξουν πρόνοιες και ρήτρε κατά της απάτης, γιατί το έχουμε δει αυτό, χωρίς να θέλω σε διανοητικό επίπεδο να τα βάλω όλα στο ίδιο καλάθι. Είδαμε στη νέα έκθεση για τη διαφθορά που έχει δώσει η Κομισιόν και που δεν μπόρεσα να την ενσωματώσω πλήρω σε αυτή την πρώτη μου έκθεση και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ίσω μέσω τροπολογιών. Έχουν εντοπιστεί χώρε αυτέ οι οποίε έχουν μεγαλύτερη φήμη και ιστορικό διαφάνειας και μη διαφθοράς, αλλά ακόμα και αυτές οι χώρες όταν βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή ε, ένωση και πηγαίνουν σε τρίτες χώρες και αυτές ξεσαλώνουν. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια μεγαλύτερη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των δράσεων των χωρών αυτών μέσω ρητρών κατά της απάτης. Εν τέλει και κλείδι θέλουμε να υπογραμμίσουμε την αναδιάρθρωση που έχει γίνει στην ΟΛΑΦ και η οποία πιστεύω ότι έχει βελτιώσει καλύτερα την συνεργασία με τα κρατη ώστε να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική διαδικασία κατά της απάτης και ιδιαίτερα στον τομέα του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων όπου βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για τη συμφωνία με τις μεγάλες επιχειρήσεις και με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουμε τη λειτουργία αυτής της συμφωνίας. Θέλω να πω τέλος ότι είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας για τα σχόλιά σας και θα προσπαθήσουμε με τις τροπολογίες σας να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή, ιδίω με τη συμπερίληψη των τελευταίων, των πιο πρόσφατων πληροφοριών που έχουμε πάρει από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ Η έκθεση είναι εξαιρετική. Πριν δώσω το λόγο να ρωτήσω κατά πόσο εκπροσωπούνται εδώ η Κομισιόν και η Όλαφ. Ε, υπάρχει δηλαδή κάποιος ε, που θα μπορούσε ή που θα επιθυμούσε να σχολιάσει τα όσα είπε μόλις η κυρία Ρέσαντερ. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κανένας. Να δώσω λοιπόν το λόγο κατευθείαν στους ε, συναδέλφους Ίγκε Γκρέσλερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν σας πω ότι αυτή η ετήσια έκθεση είναι απλώς ένα τμήμα, αν θέλετε, των πληροφοριών που διαθέτουμε όσον αφορά τις έρευνες και τα αποτελέσματα των ερευνών της όλα. Λείπει λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι από αυτό που είναι το θέμα των ορίων και έχουμε συζητήσει γι' αυτό με τον αρμόδιο επίτροπο. Δηλαδή τι σημασία έχουν αυτά τα όρια. Και αν ε, όταν θέτει προτεραιότητες διερευνητική, ο Όλαφ, τα λαμβάνει υπόψη του. Επίσης, αν τα λαμβάνει υπόψη του στην ε, στρατηγική που έχει θεσπίσει για την καταπολέμηση της απάτης και ξέρουμε ότι αυτά τα 50.000 ευρώ που ισχύουν για κάποιους άλλους τομείς, όπως παραδείγματο χάρη ο αγροτικός τομέας, αναφερόμαστε στο 1 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή οι ζημιές για τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο, αυτό μας έχει δείξει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αποτέλεσμα. 50.000 ευρώ είναι κάτι που σίγουρα δεν θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και ουσιαστικά το 99% των υποθέσεων δεν ε, αντιμετωπίστηκαν, δεν μπόρεσαν να τα επεξεργαστεί η Όλαφ καθόλου. Τελικά λοιπόν βλέπουμε ότι είχαμε στείλει και μια επιστολή τον Ιούνιο στην Όλαφ και καμία απάντηση δεν πήραμε από το Γενικό Διευθυντή. Λοιπόν, να ξέρουμε αν εδώ τι οδηγίες έχουν δοθεί από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση και βεβαίως αν μπορεί ε, η διερευνητική δραστηριότητα του Όλαφ να επεκταθεί εδώ και σε άλλους τομείς αλλά και σε ε, τι έχει να μας πει σε σχέση με τα όρια αυτά όπως έχουν θεσπιστεί. Η ερώτηση εδώ είναι πάρα πολύ ουσιαστική και σοβαρή. Έχουμε πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς εργάζεται, πώς λειτουργεί και ποια είναι η αποτελεσματικότητα του Όλαφ εδώ. Έχουμε λοιπόν κάποιες εσωτερικές, ε, όπως τις λένε, έρευνες, οι οποίες είναι αποκλειστική αδερμοδιότητα του οργανισμού και γι' αυτό πρέπει να πω ότι θα ήθελα εδώ να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου. Οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν. Ο Επίτροπος Έμετα μας απάντησε γραπτά λέγοντας ότι δεν ισχύει αυτή η ερώτηση. Για μας αυτή η ερώτηση είναι ουσιαστική για την καθημερινή λειτουργία και δραστηριότητα του Όλαφ και πραγματικά είναι θέμα στρατηγικής και είναι κάτι που καθορίζει πραγματικά την καθημερινή εργασία και δραστηριότητα αυτού του οργανισμού. Δεν βλέπω λοιπόν κάποιον από την Επιτροπή εδώ, ελπίζω να μας ενημερώσουν ε, με τη γραπτή διαδικασία. Πώς λειτουργεί, επαναλαμβάνω, Όλαφ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση και το υπογραμμίζω και το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παραδείγματο χάρη, και της αλληλεπίδρασης ε, με αυτά που κάνει όλα αυτά. Το πώς θα καταπολεμήσουμε την απάτη, μα είναι κάτι που μας απασχολεί και μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στους τομείς που έχουμε εντοπίσει, είναι ένα κεφάλαιο. Από την άλλη, η φοροεισπρακτική ικανότητα, η δυνατότητα να συγκεντρωθούν έσοδα. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι το θέμα των ορίων δεν αναφέρεται καθόλου στην έκθεση. Θα θέλαμε λοιπόν εδώ κάποιες απαντήσεις και κάποια άλλα σημεία για τα οποία χρειάζεται πιο συγκεκριμένη απάντηση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η τελευταία έκθεση PIF δεν έχει επεξεργαστεί, δεν την έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες αγνοήθηκαν. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η προηγούμενη έκθεση δεν έχει καν γίνει αντικείμενο επεξεργαστή, ίσως θα έπρεπε να μην προετοιμάσουμε τη νέα έκθεση. Είμαστε υπομονητικοί, αλλά δεν είναι δυνατόν εδώ να μην υπάρξει μία ανταλλαγή απόψεων, μία αντιπαράθεση η οποία θα οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ε, άλλες παρεμβάσεις. Ζητάει κάποιος άλλος το λόγο. Κυρία Γιάλα. Θέλετε το λόγο, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι Ίγκεμπορκ ότι δεν έχω αυτή την πληροφορία τελευταία στιγμή σε σχέση με την ΟΛΑΦ. Ε, Εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορείς να κάνεις αυτό το οποίο λες και θα σε υποστηρίξω κάτι άλλο. Θέλω να τονίσω ότι πάντα έχουμε αντιμετωπίσει την ε, απάτη για τα θέματα δαπανών. Και επειδή ο προπολογισμό μα είναι όλο και μικρότερο, θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο και για, τις, ε, για τα έσοδα του προπολογισμού. Δεν μιλάω για την Όλαφ, μιλάω για την απάτη που γίνεται στα έσοδα τη ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό έχω τονίσει τα θέματα του, της απάτης στο ΦΠΑ και την καλύτερη παρακολούθηση των θεμάτων αυτών στον τομέα και των εσόδων και των ε, δαπανών. Συμφωνώ λοιπόν για την ε, Όλαφ ότι πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες ενέργειες. Πρέπει να έχουμε καλύτερη εποπτεία της Όλαφ, αλλά από τη στιγμή που θα υπάρξει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, αυτό είναι πια ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κάνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας και εδώ θα είναι πολύ μικρός ο χώρος των κρατών μελών που δεν θα δεχτούν την ύπαρξη και τον έλεγχο από την πλευρά του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Νομίζω ότι δημιουργούμε έτσι ένα πλαίσιο ποινικού δικαίου που θα είναι σαφές και θα έχουμε σαφείς κανόνες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την δίωξη των ε, αδικημάτων στον τομέα αυτό και ελπίζω θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε και Έχουμε και εμείς λάβει σαν βάση την έκθεση του Derek και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε λοιπόν σε μια πιο πλήρη αντιμετώπιση της κατάστασης της εφαρμογής του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και μια καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος για το γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις της Κομισιόν ή του Κοινοβουλίου. Και είμαι έτοιμη λοιπόν να δεχτώ τις τροπολογίες σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ανακοινώνω τις προθεσμίες για τις τροπολογίες 22 ε, Φεβρουαρίου του 2014, 12 η ώρα το μεσημέρι. Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας ε, συνεδρίαση, η ημερήσια διάταξη του πρωινού. Να σας ενημερώσω Sorry. Következő alkalommal módunk lesz majd a kont képviselőivel erről a kérdésről. E- Την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να επανέλθουμε ε, στην ανταλλαγή απόψεων ε, επί του θέματος με τα μέλη της Επιτροπής Κοντ 20 Φεβρουαρίου. Από τις 9 η ώρα είναι η επόμενη μας συνεδρίαση. Θα πρόκειται για εκείνη η συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχετε τον λόγο, κυρία Σανδεύ. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά είπατε ότι είναι το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου, προθεσμα για τις τροπολογίες. Α, 25, δεν σας άκουσα καλά. Συγγνώμη, γιατί 22 ήταν Σάββατο. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους, επειδή έχει έρθει η εκπρόσωπος του, της ΟΛΑΦ εδώ, έχουμε κλείσει κανονικά τις εργασίες μας, αλλά επειδή είχαν τεθεί ορισμένα ερωτήματα μήπως θέλετε να δώσουμε τη δυνατότητα στην εκπρόσωπο της ΟΛΑΦ να λάβει το λόγο για την έκθεση για την προστασία των ε, ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήσεις και να αναφέρουμε τις ε, ανησυχίες μας σε σχέση με τις τιμές κατοφλίου πρώτα απ' όλα και δεύτερον σε σχέση με τις προτεραιότητες για το 2014 όπου οι δαπάνες βρίσκονται σε τέταρτη θέση. Εγώ θα προβλεπόταν να ε, κάνω την εξέταση του σημείου μου στις 12. Αν θέλει λοιπόν η Όλαφ μπορεί να μας δώσει ορισμένε διευκρινήσει για τα θέματα αυτά. Αν θέλει. Καλό δεκτή είναι πάντα η, η αξιολόγηση αυτή. Εγώ δεν θέλω να ξαναλέω δύο και τρεις φορές την ίδια ιστορία. Δεν είναι τρόπος ε, λειτουργίας αυτό μιας ε, επιτροπής. Συνάδελφοι, συμφωνώ και εγώ. Εγώ μου είχαν πει ότι θα λάβω το λόγο. Μου είχαν πει ότι θα λάβω το λόγο στις 12 και φαντάζομαι ότι και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και της ΟΛΑΦ προβλέπαν να κάνουν τη συζήτηση αυτή στις 12. Εγώ νομίζω ότι έχουμε ακόμα λίγο χρόνο και εγώ θα ήθελα να ακούσω, αν δεν θέλει κανένα άλλος, την άποψη της ΟΛΑΦ και της Κομισιόν. Παρακαλώ. Tisztelt képviselőtársaim, mielőtt bonyolult ügyrendi vitába bocsátkoznánk. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω λοιπόν να δώσουμε αμέσω το λόγο στους εκπροσώπους της ΟΛΑΦ, χωρίς άλλα διαδικαστικά. Δεν είναι λάθος τους, ήρθαν λίγο καθυστερημένα. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να μας πούν τις απόψεις τους. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να, να σας πω ότι ήρθαμε λίγο καθυστερημένα, αλλά θεωρούσαμε, όπως είπε και η συγγήτρια, ότι αυτό το σημείο θα συζητηθεί στις 12. Λυπούμεθα πολύ λοιπόν, γιατί δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε μέχρι τώρα την συζήτηση. Κυρία Γκρέσλε, δεν άκουσα την ερώτησή σας αλλά βεβαίως ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου καταρχήν ε, γενικά να αναφερθώ στο σχέδιο έκθεσης της κυρίας ε, Αγιάλα. Η Επιτροπή θα ήθελα να πω ότι εκπλήσεται πολύ ευχάριστα από την πολύ ισορροπημένη έκθεση και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Συνήθως εργαζόμαστε αγγλικά ή γαλλικά. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι πρόκειται για μια πολύ ισορροπημένη και οικοδομητική έκθεση και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Είναι ένα πολύ θετικό σημάδι εν των ευρωπαϊκών εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της απάτης που πλήττει τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Στην έκθεση αυτή λοιπόν υπάρχουν ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Οδηγία ΠΙΦ, πρωτοβουλία ΕΠΟ που ψηφίστηκε σήμερα το πρωί εδώ και βεβαίως η μεταρρύθμιση που θα η μεταρρύθμιση του Όλαφ που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013. Πέρσι η ανακοίνωση για τα τσιγάρα, το πρωτόκολλο CTC, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης που πλήττουν τον κοινοτικό προπολογισμό περιέχουν λοιπόν όλες αυτές τις προτάσεις, τις δράσεις. Θυμάστε μάλιστα την οδηγία για τις κρατικές, τις δημόσιες προμήθειες που υιοθετήθηκε και που οδηγεί σε περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις κρατικές, τις δημόσιες προμήθειες. Πολύ σημαντικό βήμα και αυτό. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος μεν, παρόλα αυτά οι προσπάθειές μας θα πρέπει να συνεχιστούν. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη-μέλη, γιατί όπως γνωρίζετε η ευθύνη των κρατών μελών είναι μεγάλη στην καταπολέμηση της απάτης. Ο κανονισμός που αφορά τον Όλαφ συμπεριλαμβάνει δράση από μέρους των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη. Σήμερα υπάρχουν υπηρεσίες για την καταπολέμηση της απάτης σε όλα τα κράτη-μέλη και βεβαίως πρέπει να γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και μία αναφορά πλέον γίνεται δεσμευτικό αυτό στην, ε, από τα κράτη-μέλη μέσω αυτής της υπηρεσίας των Όλαφ. Οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Budget με ενημερώνουν ότι υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν τις προτεραιότητες επενδύσεων αλλά και το θέμα των ορίων των κατόφλιων. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσω βεβαίως ε, με πολλές λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι ο κανονισμός 88.3 που θα ζητηθεί τον Απρίλιο μεταξύ των θεσμικών οργάνων με παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Όλαφ καθώς και της ε, Επιτροπής Εποπτείας θα ολοκληρωθεί κανονικά τέλος Απριλίου. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα σημεία που θα συζητηθούν, θα εξεταστούν, όπως οι προτεραιότητες για τις έρευνες, τις διερευνητικές διαδικασίες της Όλαφ, του Όλαφ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρέσλε. Δεν ήθελα να λάβω το λόγο, αλλά σήμερα κανείς δεν φαίνεται να είναι προετοιμασμένος για τα ερωτήματα αυτά. Για το θέμα του και για τα κατόφλια. Λυπάμαι που φαίνεται ότι εψεύστη προς εμάς η Κομισιόν. Και οι προτεραιότητες, τι ρόλο παίζουν οι προτεραιότητες στο έργο της ΟΛΑΦ. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε για τα κατόφλια που φαίνεται ότι μερικές φορές είναι το μοναδικό κριτήριο που χρησιμοποιείται για δράση από την πλευρά της ε, ε, βλέπω ότι και από την έκθεση του 2012 υπάρχουν ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Και αν τελικά κάνουμε συνεδρία σε επιτροπής και όλα τα στοιχεία δίνονται έγγραφα στη συνέχεια και δεν δίνει κανείς πληροφορίες προφορικά, τι νόημα έχει να κάνουν αυτές οι συνεδριάσεις επιτροπών. Τι νόημα έχει να κάνουμε λοιπόν αυτά τα κατόφλια θα ήθελα να ξέρω στο ρόλο, στο έργο της ε, Όλαφ, τι έκαναν το 2012, τι γίνεται με τις εσωτερικές έρευνες οι οποίες ποτέ δεν έχουν ε, αναδυθεί ως ε, προτεραιότητα παρά το γεγονός ότι είναι μέσα στην αρμοδιότητα της Όλαφ και τι γίνεται για όλες αυτές τις περιπτώσεις που βρίσκονται κάτω από το κατόφλι. Τι μπορούμε να ξέρουμε για τη συνέχεια που δόθηκε για τα θέματα αυτά. Μήπως θα μπορούσε η Όλαφ να μας δώσει πληροφορίες πιο σύντομα να μειωθούν τα χρονικά δια, ε, όρια για την πληροφόρηση. Αναφερθήκατε στα, στα θέματα το, της αγροτικής ε, ανάπτυξης αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις που αντιμετώπισε η Όλαφ δεν εμπλέκονται σε αυτά τα κατόφια. κατόφια. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να έχουμε απαντήσει όλα αυτά τα θεματα ehm, Υπάρχουν άλλα σχόλια, ερωτήσεις, ε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Αν όχι, να δώσω ξανά το λόγο στην εκπρόσωπο της ΟΛΑΦ. Σας ευχαριστώ. Ζητώ την κατανόησή σας. Γιατί δεν μπορώ να μπω τώρα στις λεπτομέρειες των ερωτήσεων της κυρίας Κρέσλε. Θέλω όμως να το τονίσω ότι αυτό γίνεται ότι θα πρέπει να ακούσετε την άποψη της Γενικής Διεύθυνσης. 8 Απριλίου αναφέρθηκαν οι προτεραιότητες για το 2014. Αυτό είναι ένα σημείο που θα συζητηθεί λοιπόν στη συνέχεια και δεν μπορώ εγώ τώρα να το προκαταλάβω. Για τις προτεραιότητες του 2013 ξέρω ότι έλαβαν χώρα κάποιες συζητήσεις και συζητήθηκαν τα θέματα αυτά και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Το 99,8 που ανέφερε η κυρία Γκρέσλε το λαμβάνω υπόψη, αλλά νομίζω ότι η κυρία Γκρέσλε σε μια συνάντηση είχε τονίσει ότι μόνο ένα πολύ περιορισμένο ποσοστό περιπτώσεων δεν αντιμετωπίστηκε και τα κατόφλια δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο σε κάτι τέτοιο. Το 2014 δεν έχουμε πια τέτοια κατόφλια σε σχέση με τα ποσά πληρωμών, αυτό που θέλω να το τονίσω και κατά τα άλλα είναι σαφής η άποψή μας σε σχέση με τις ε, ανακρίσεις, τις έρευνες. Ακολουθούμε τη διαδικασία του άρθρου 5 και όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις αυτού του άρθρου, εμείς ξεκινάμε αυτές τις ε, ε, έρευνες. Παραθέτω επίσης αυτό το οποίο λέγεται ότι η απόφαση έναρξης ερευνών λαμβάνει υπόψη της προτεραιότητος και την πολιτική του γραφείου που θα λάβει υπόψη την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματική χρήση των πόρων του γραφείου της ΟΛΑΦ δηλαδή και αναλογικότητα σε σχέση με την ε, ανάγκη αντιμετώπισης σε επίπεδο ερευνών. 8 Απριλίου λοιπόν ο κύριος Κέσλερ θα σας δώσει πιο πολλές λεπτομέρειες για όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Ναι. Κοιτάξτε, τι να σας πω. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η στρατηγική καταπολέμηση της απάτης της Επιτροπής και υπάρχουν κάποια κριτήρια. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι τι νόημα, τι ρόλο παίζουν αυτά τα όρια, τα κατόφλια για την εργασία και τις επιλογές του Όλαφ. Εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο καθότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προστατευθούν. Έχω κάνει μια ολόκληρη, αν θέλετε, ε, προσπάθεια να στοιχειοδοτήσω και να δικαιολογήσω την ε, θέση μου και βασίζεται σε αυτό. Πριν τις 8 Απριλίου δεν μπορείτε να μας απαντήσετε. Γιατί εμείς για το 2012 έχουμε μία προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Απαντήστε μας και για την ΠΙΦ, αλλά και για το θέμα της Όλαφ. Σας ευχαριστώ πολύ αν το κάνετε. Είπατε ότι η έκθεση είναι πολύ ισορροπημένη, αλλά πραγματικά, ναι, υπάρχει γραπτή διαδικασία, θα τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά υπάρχει και προφορική. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Γκάιερ. Λοιπόν, ακούσαμε το θέμα των τροπολογιών, της προθεσμίας για την έκθεση Αγιάλα. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Γκέ Γκρέσλε. Τώρα, όσον αφορά τα όρια όμως, τα κατόφλια, τις τιμές, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει θίξει το θέμα αυτό και συμφωνώ ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε με τον Επίτροπο. Αν ακολουθήσουμε την δική σου τοποθέτηση ότι το 99, κάτι των υποθέσεων δεν τις αντιμετωπίζει η καθόλου Όλαφ, τελικά παραμένουν ελάχιστα, αν θέλετε, ιδιαίτερα παραδείγματος χάρη στον τομέα το γεωργικό. Και ουσιαστικά βλέπουμε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις ε, απάτης δεν, επεξεργα... δεν μπορεί να τις επεξεργαστεί καθόλου Όλαφ και σε άλλους τομείς. Η σημασία λοιπόν αυτών των ορίων, κατά την άποψή μου, βέβαια παίζουν ένα ρόλο όσον αφορά την επιλογή των υποθέσεων από τον Όλαφ. Ποιες υποθέσεις θα ε, επιλέξει, αλλά είναι ένα από τα κριτήρια. Δεν είναι το καθοριστικό κριτήριο και το μοναδικό κριτήριο. Μπορεί η Επιτροπή να μας δώσει και κάποιες άλλες εξηγήσεις, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι η καταπολέμηση της απάτης, ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, δεν βασίζεται μόνο σε αυτό το κριτήριο, αν θέλετε, των ε, ορίων αυτών. Η κυρία Γκρέσλε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το νούμερο αυτό δεν τον έβγαλα από το μυαλό μου. Η Γενική Διεύθυνση για την ε, Γεωργία την, τώρα έχει υπολογίσει αυτό. Και είναι του Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου του 2013. Η Γενική Διεύθυνση μας είχε μιλήσει για αυτήν την υπόθεση λέγοντας ότι όντως, όπως ξέρετε είναι ακόμα πιο ψηλό το όριο για τη γεωργία και ότι πραγματικά ένα ελάχιστο ποσοστό των υποθέσεων φτάνουν μέχρι τον Όλαφ για επεξεργασία. Αυτό πραγματικά ε, είναι κάτι που μας ανησυχεί. Δηλαδή, ποιος επιλέγει. Γιατί ιδρύσαμε τον Όλαφ. Γιατί κάποιες υποθέσεις δεν διαλευκανόταν και δεν ασχολόταν τα κράτη-μέλη μαζί τους. Αν δεν τις ε, αναλαμβάνει αυτές τις υποθέσεις ούτε ο Όλοφ, μα τότε έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα και προσπαθώ εδώ να πω ότι πάρα πολλές τέτοιες ε, υποθέσεις καταπολέμησης της απάτης που είναι γνωστές αν θέλετε. Δεν τις επεξεργάζεται κανείς και πραγματικά εγώ θα ήθελα εδώ να επιστήσω την προσοχή σας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν βλέπω, δεν είμαι αποσιόδοξη και δεν βλέπω το ποτήρι μίσο άδειο. Επαναλαμβάνω, πάνω από 99% των υποθέσεων δεν είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τον Όλαφ. Κύριε Γκρέσλε, προφανώς θα το εξετάσω αυτό το θέμα, μα ξέρω και εγώ προσωπικά αυτά τα θέματα που αναφέρατε από τη Γενική Διεύθυνση για τα Αγροτικά Θέματα τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2013, ό,τι δεν ξέρω προφανώς θα το ερευνήσω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορώ να δω τις στατιστικές μας για το 2012 και για τις εκθέσεις του 2013 και ο κύριος Κέσσερ θα σας πει στις 8 Απριλίου και τα τελευταία στοιχεία και είναι σαφές ότι εμείς ε, επεξεργαζόμαστε περισσότερες και όχι λιγότερες περιπτώσεις. Και πράγματι εξετάζουμε μέσα στα, ό,τι μπορούμε μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μας. Θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι σε όλους τους τομείς, ακόμα και την αγροτική ανάπτυξη, εμείς είμαστε ιδιαίτερα ενεργοί. Θα εξετάσω λοιπόν αυτά που αναφέρετε, αλλά νομίζω ότι και αυτά τα οποία ισχύουν για την αγροτική ανάπτυξη είμαστε πάρα πολύ ε, ενεργοί και για το 2015 οι προτεραιότητές μας θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ε, ενεργητικότητα. Τα κατόφλια δεν ήταν λοιπόν ε, προϋποθέσεις δράσης ή όχι. Ήταν κάτι που συνεκτιμούσαμε στην συνολική εικόνα για την δυνατότητα δράσης μας και επομένως τα νέα, οι νέες προτεραιότητες μας δεν αναφέρουν καθόλου κατόφλι. Από ό,τι γνωρίζω λοιπόν, για τα στοιχεία του 2012-2013. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, αλλά θα ξε, ξαναερευνήσω τα στοιχεία αυτά. Κυρία Γκρέσλε. Λυπούμε, λυπούμε. Θα λέω για τρίτη φορά. 2012, για το 2012 έχουμε πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία. Τι να σας πω, θα σας προετοιμάσω και μια γραπτή ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση. Δεν είναι δυνατόν ε, πλέον με τόσες πολλές στατιστικές να συγκρίνει κανείς το τι υπήρξε πριν και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πάνω από 400.000 υποθέσεις Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι πάρα πολλά. Τι είναι λοιπόν εδώ αξιόπιστο, πώς μπορούμε να βασιστούμε σε συγκρίσιμα στοιχεία και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι μειώνεται η αποτελεσματικότητα του Όλαφ. Αν δει κανείς ποια είναι τα σημεία, ποιες είναι οι υποθέσεις που αποφάσισε να διερευνήσει ο Όλαφ, αν παρακολουθήσουμε αυτές, το 20% αυτών δεν μόνον οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα. Ούτε καν το 50%. Και μπορώ να σας δείξω αυτά που σας λέω με τις στατιστικές που διαθέτουμε. Αυτό προσπάθησα να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω, επαναλαμβάνω, νούμερα και στοιχεία τα οποία να είναι συγκρίσιμα. Αλλά πολλές φορές είναι αδύνατον. Γιατί η αλλαγή, η μεταρρύθμιση στον Όλαφ δυστυχώς μας οδήγησε σε μια κατάσταση που δεν είναι πλέον εύκολο να συγκριθεί σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς και να μην κρύβουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανταλλαγή Απόψε Θα δώσω για άλλη μια φορά το λόγο στην εκπρόσωπο του ΟΛΑΦ και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Γιάλα Σαντέρ για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της ημερησής δίδαξης για δεύτερη φορά. Σας ευχαριστώ. Μου ξαναδίνετε το λόγο και πάλι. Και να πω στην κυρία Γκρέσλε, έχετε δίκιο, γιατί το 2012 είχαμε αλλάξει την, ε, τις στατιστικές μας, γιατί αυτό οφείλεται στην μεταβολή της ε, δομής της Όλαφ, είχε συζητηθεί αυτό το θέμα, τον Φεβρουάριο του 2012 είχε αλλάξει η δομή της Όλαφ και οι διαδικασίες έρευνας είχαν προσαρμοστεί για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της Όλαφ. Γι' αυτό το 2012 ήταν ένα έτος μετάβασης και αυτό αντανακλάται στην έκθεση της ε, όλα, Αλλά το κάναμε αυτό πάρα πολύ σαφές και το ανακοινώσαμε με απόλυτη διαφάνεια και φυσικά μια γενική διεύθυνση πάντα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην οργανωτική δομή που κατά την άποψή μας οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ερευνητικών μας διαδικασιών. Και σας λέω και πάλι, στις 8 Απριλίου θα παρουσιαστεί η έκθεση του 2013 και σας τονίζω ότι τα αποτελέσματα μας ήταν πολύ καλά. Αυτό δείχνει ότι ήταν αποτελεσματικές και επωφελείς οι αλλαγές <clears throat> που έγιναν ε, το 2012. Και αυτά θα φανούν στην έκθεση που θα δημοσιεύσουμε τον Απρίλιο. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Άγια Λασέντερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι μπόρεσα να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση για να τη λάβω υπόψη σε σχέση με τις τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν. Εγώ θέλω να πω και πάλι ότι το θέμα αυτό των ε, αριθμών είναι πολύπλοκο και μπορεί ο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία υπέρ ή μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κατά. Αλλά όταν αλλάζουν τα στοιχεία και για το και από το ελεγκτικό συνέδριο, δεν είναι εύκολο να εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία αυτά. Δεν πρέπει να είμαστε λοιπόν μεροληπτικοί για τα στοιχεία όταν είναι καλά να θεωρούμε ότι δεν είναι καλά επειδή άλλαξαν και όταν είναι κακά να θεωρούμε ότι μπορεί να μην είναι κακά επειδή προέρχονται από μια αλλαγή. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια προς το παρόν τουλάχιστον λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Εν πάση περιπτώσει κατανοώ ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή στο έργο της ΟΛΑΦ. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στην ΟΛΑΦ για να υπάρξουν θετικότερες ε, αλλαγές. Όταν τώρα έχουμε όμως μία επιστολή για τα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης που οδηγεί σε βαριές κατηγορίες και όταν εμείς αλλάξαμε το σύστημα για την αγροτική ανάπτυξη με τη συγχρηματοδότηση. Όλα αυτά δεν μας δίνουν τη δυνατότητα ούτε να κατηγορήσουμε την Γενική Διεύθυνση για τα αγροτικά θέματα, ούτε για να θεωρήσουμε ότι φταίει σε αυτά η όλα. Εδώ έχουμε το ελεκτικό συνέδριο που είπε ότι οι αποτελέσματα αυτής της αλλαγής ήταν αρνητικά γιατί άλλαξε ο μηχανισμός ελέγχου και επήλθε η διαδικασία συγχρηματοδότηση με τα κράτη-μέλη. Τώρα το αν αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά θα πρέπει να ερευνήσει τέτοιε περιπτώσει. Η κυρία Χόφμαν είπε σωστά ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιε ενδείξει για να προβεί η Όλαφ σε ελέγχου. Εγώ θα ήθελα να ήταν εδώ ο Γενικός Διευθυντής της, ε, της ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας να μας δώσει πληροφόρηση που θα ήταν σαφής και διάφανη για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Δεν μπορώ εγώ να ψάχνω τον κάθε Γενικό Διευθυντή. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η επιστολή και θέτει το βάρος στους ώμους της όλα, θα θέλαμε να είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτά που λέει ο Γενικός Διευθυντής της, ε, της Άγκρη. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε όλοι τις πληροφορίες αυτές και να μπορέσουμε να συζητήσουμε εν γνώση της κατάστασης. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι θέμα μονάχα μαζί μου να είναι εντάξει, αλλά η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, αλλά πρέπει όλοι οι, οι να ξέρουν αν έχει αλλάξει γνώμη ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής Γεωργίας και αν υποστηρίζει την ΟΛΑΦ ή όχι και να μην χρειάζεται να ψάχνουμε δεξιά και αριστερά για να δούμε τελικά ποιος είναι ο υπεύθυνο για αυτά τα πράγματα και πού πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, για τις τροπολογίες. Προθεσμία είναι 12 το μεσημέρι στις 25 Φεβρουαρίου και όπως είπα ήδη 20 Φεβρουαρίου στις 9 η ώρα θα έχουμε την επόμενη μας συνεδρίαση από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έτσι θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Εδώ ολοκληρώνεται συνεδρίαση. Ευχαριστώ.